Καλώς ορίσατε στη συνεδρίασή μας. Στην πρώτη μας συνεδρίαση συγκεκριμένα. Την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια είχαμε μια από κοινού συνάντηση για μια μισή ώρα με άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. Τώρα ξεκινάμε τις δικές μας διαδικασίες. Ελπίζω ότι περάσατε καλά στις διακοπές σας και είστε ευτυχείς με την επιστροφή σας εδώ. Σε μία ώρα θα έχουμε και ψηφοφορίες, σε μία ώρα. Τώρα για την ημερήσια διάταξη δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια σχόλια, μπορεί να γίνει δεκτή η ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Για τις ανακοινώσεις από πλευράς μου δεν έχω να σας μεταφέρω κάτι ιδιαίτερο σήμερα. Αν υπάρξει κάτι, αν παρουσιαστεί κάτι ε, πριν τις ψηφοφορίες θα σας το μεταφέρω. Πηγαίνουμε τώρα στο σημείο 3, έγκριση πρακτικών. Αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις για τη συνεδρίαση 18 και 19 Ιουνίου. Το σημείο 4 τώρα Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή, προκλήσεις, ευκαιρίες και μαθήματα για τη σχεδίαση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η συγητής μας εδώ είναι ο συνάδελφος Τάμας Ντότς. Δυστυχώς όμως ο εισηγητής δεν μπορεί να είναι σήμερα μεταξύ μας γιατί καθυστέρησε πάρα πολύ η πτήση του. Θα έρθει, αλλά θα έρθει αργότερα. Και γι' αυτό ο κ. Ντέλη θα τον αντικαταστήσει. Υπάρχουν και οι σκιώδεις που μπορούν να πάρουν το λόγο μετά. θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Γι' αυτό ο Αντόρ Ντελή του ζητώ να μας παρουσιάσει τις θέσεις του εισηγητή. Εγώ απλά θα σας μεταφέρω τις σημειώσεις του κύριου Ντότς για την πρότασή του και θα συνεχίσω στην Ουγγρική. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης είναι κάτι το απαραίτητο πλέον, έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκμεταλλευτεί την κατάσταση αυτή. Όπως λέει και το πρόγραμμα δράσης, υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες στην ψηφιοποίηση που θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε ε, την εκπαίδευση. Ο διεθνής ανταγωνισμός αυξάνεται και σε επίπεδο χωρικό και σε επίπεδο χρονικό. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Στόχος των εκπαιδευτικών συστημάτων είναι η βελτίωση των ανθρώπινων πόρων, των ανθρώπινων ικανοτήτων και η προετοιμασία των φοιτητών και διαμέσου της διαβίου κατάρτισης να προσαρμόζονται στις νέες αλλαγές με υψηλές ταχύτητες. Πρέπει να σας ενθαρρύνω όλους να συμμετέχετε πλήρως, να ενθαρρύνουμε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν πλήρως στις διαδικασίες της ψηφιοποίησης. Με δύο τρόπους επηρεάζεται η εκπαίδευση. Καταρχάς οι πολίτες οι οποίοι φεύγουν από τον χώρο της εργασίας πρέπει να προετοιμάζονται σωστά και για να επιστρέψουν. Και δεύτερον, οι ψηφιακές τροποποιήσεις θα πρέπει στο εσωτερικό των τακτικών, θα έλεγα, εκπαιδευτικών διαδικασιών να αποκτήσουν βαθύτερη, ε, βαθύτερες ρίζες και όπως σας είπα και στην αρχή της παρουσίασής μου, όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούν ψηφιακές γνώσεις. Συνεπώς ε, θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι γνώσεις αυτές μπορεί να προστιθένται. Θα απαιτηθεί ένα ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων και όλοι οι πολίτες που ολοκληρώνουν κάποια επίπεδα εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν αυτά τα ε, προαπαιτούμενα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει, ε, θα έλεγα, στροφή στην λεγόμενη κάλυψη των προσωπικών αναγκών των σπουδαστών και γι' αυτό και στον ψηφιακό επίπεδο θα πρέπει να βελτιώσουμε την δικαιοσύνη και την αποτελεσματικότητα οι οποίες θα πρέπει να διέπουν την εκπαίδευση θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε σωστά φυσικά και τους διδάσκοντες. Αυτό θα πρέπει να γίνει με συστηματικό τρόπο και να πω εδώ ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και οι καινοτόμες δράσεις στον τομέα των ψηφιακών απαιτούν ψηφιακές δράσεις υψηλής ταχύτητας. Γι' λοιπόν αυτό και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι επενδύσει στον τομέα τη εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά τώρα το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, πρέπει να δημιουργηθούν εταιρικέ σχέσεις και να διατηρηθούν ήδη φυστάμενε. διότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βελτιώσουμε και τις συνθήκες διαβίωσης στην κοινωνία. Επίσης, ο εισηγητής ε, στο τέλος ε, του σημειώματος αναφέρει πως ε, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν δεν μπόρεσε να συμπεριλάβει όλες τις σκέψεις. Θα καταθέσει λοιπόν τροπολογίες σε συνεχεία. Προσβλέπει βέβαια και στη συμμετοχή των συναδέλφων ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε συνάδελφε για τη βοήθειά σας, για την παρουσίαση και περνάμε στους σκιώδεις εισηγητές. Εκ μέρους ε, Σοσιαλιστών Δημοκρατών, ο κύριος Ζωρίνο θα αντικαταστήσει συνάδελφο που έπρεπε να είναι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η σκιώδης ήτρα δεν μπορούσε να είναι εδώ. Μου ζήτησε όμως να παρουσιάσω εγώ εκ μέρους της τη θέση της ομάδας μας, την οποία και συμμερίζομαι. Καταρχάς, ε, ένα ευχαριστώ προς τον εισηγητή για τη δουλειά του. Θεωρούμε πως έχει εστιάσει σωστά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε καλή ανακοίνωση, σε καλές ανακοινώσεις σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά και το συγκεκριμένο θέμα που μας απασχολεί είναι σημαντικό. Για το μέλλον οι ψηφιακές τεχνολογίες θα προσλάβουν ακόμα μεγαλύτερη ε, σήμαση για την καθημερινότητα και την επαγγελματική ζωή των συμπολιτών μας. Θα πρέπει λοιπόν ε, τα νέα ψηφιακά πρότυπα, οι ψηφιακή ψηφιακοί κανόνες να μπορέσουν να εσωματωθούν. Θα πρέπει να υπάρχει η πρόσβαση σε όλους ε, και ιδίως μιλώ για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας που θεωρούν ότι αποκλείονται ή δεν μπορούν να συμμετέχουν. Οι δεξιότητες, η κατάρτιση είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ψηφιακή εποχή. Όσοι εργαζόμενοι δεν έχουν τέτοιου είδους γνώσεις μέχρι στιγμής θα πρέπει να καλύψουν το κενό αυτό για να μην μείνουν πίσω. Δεν θέλουμε ούτε διακριτική μεταχείριση ούτε εμπόδια φραγμούς λόγω ηλικίας ή φύλου. Εξού και αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση για όλους και σε μία δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση. Η ψηφιακή ε, διδασκαλία, η ψηφιακή εκμάθηση είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλους. Όλοι πρέπει να αποκτήσουμε τις απαραίτητες αυτές δεξιότητες και ικανότητες. Αυτό είναι κάτι που το χρειάζονται όλοι, και τα παιδιά μας και ο κύκλος μας γενικώς. Υπάρχει κάτι τώρα το οποίο μου φαίνεται κάπως περίεργο σε ό,τι αφορά τη γνωμοδότηση. Δεν είναι ακόμη γνωστή η έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας Επιτροπής Πολιτισμού. Και πάνω σε αυτήν ουσιαστικά εμείς ε, καταρτίζουμε μια γνωμοδότηση. Δύο ημέρες μένουν για τη λήξη προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών. Είναι κάπως περίεργη αυτή η διαδικασία. Περιμένουμε και ελπίζουμε η δική μας γνωμοδότηση να συμπεριληφθεί στην ε, έκθεση που συντάσσει η Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Αλφα, για την παρουσίαση αυτή. Μέρος της Άλντε, η κυρία Πόνσετς, που δεν είναι εδώ. Η κυρία Νάρτιγκέλ θα την αντικαταστήσει. Um, Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Δυστυχώς, η κυρία Πότζεκ δεν είναι εδώ. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω τα ακόλουθα. Το πρώτο σημείο που θέλω να πω είναι ότι ο, ο κόσμος αλλάζει γρηγορότερα από ποτέ. Και οι ψηφιακές αλλαγές είναι πραγματικά επαναστατικές ε, σε όλους τους τομείς. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν το περιβάλλον εργασίας με τρόπους που ποτέ δεν είχαμε φανταστεί. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η εκπαίδευση και η κατάρτιση γίνονται όλο ένα και πιο σημαντικές στην ε, κατάρτιση όλων των εργαζομένων. Συμφωνούμε με τον εισηγητή ε, σε ό,τι αφορά την θέση του ότι η κατάρτιση είναι η πιο σοφή επένδυση για το μέλλον. Η ψηφιακή τεχνολογία εμπλουτίζει την εκπαίδευση με όλες αυτές τις ευκαιρίες εκμάθησης αλλά και ευρείας, και μιας ευρείας γκάμας ερευνητικών εργαλείων. Η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει την καινοτομία στην εκπαίδευση. Τα ανοιχτά δεδομένα δεν είναι μόνο ερευνητικό εργαλείο, αλλά και ένα εργαλείο ανάπτυξη σε διάφορους επιστημονικούς τομείς. Η πρόσβαση όμως σε όλες αυτές τις ευκαιρίες εξαρτώνται από την υποδομή και απαιτούν υψηλού επίπεδου συνδεσιμότητα. Η σημασία λοιπόν αυτής της συνδεσιμότητας και του να υπάρχει η υποδομή για όλα αυτά τα ταχεία δίκτυα θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την απασχόληση. Η... Είναι ανάγκη να ενδυναμώσουμε αυτού του τύπου τις ευκαιρίες εκμάθησης, αλλά και ψηφιακές ευκαιρίες και πρωτοβουλίες που συμπεριλαμβάνονται και στο πρόγραμμα 2020, ούτω ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε συγκεκριμένες δεξιότητες. Υπάρχει επίσης και η ανάγκη να ενδυναμώσουμε τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Και στα πλαίσια αυτά της έρευνας και καινοτομία με τις διάφορες κοινότητες, οι διάφορες κοινότητες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Θέλουμε επίσης να δώσουμε σημασία και στα διάφορα πιλωτικά προγράμματα σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Θα πρέπει να κρατάμε κατά νου το ανθρώπινο δυναμικό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ευρωπαϊκές οικονομίες και αυτές οι ψηφιακές δεξιότητες δεν είναι πλέον μια πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχει κάποιος που θέλει να προσθέσει κάτι. Όχι. Εκ μέρους των Πρασίνων τώρα. Ο Μπένεντικ Γιάβολ έχει το λόγο. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και τον εισηγητή. Θέλω απλώς να αναφέρω τέσσερα επιπλέον ζητήματα που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά την προσαρμογή μας στην ψηφιακή κοινωνία. Πρώτα απ' όλα, την ανάγκη της εκπαιδευτικής στήριξης στο ε, επαγγελματικό περιβάλλον, ώστε να μπορέσει να γίνει αυτή η μετάβαση καθώς η αγορά εργασίας αλλάζει ταχύτατα, όπως ανέφερε και ο εισηγητής, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να προσφέρουμε την απαιτούμενη στήριξη στους εργαζόμενους, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε αυτή την ψηφιακή αγορά εργασίας. Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να θίξω είναι η ίση πρόσβαση στις ψηφιακές ευκαιρίες. Πράγμα το οποίο δεν σημαίνει απλά τεχνική πρόσβαση. Υπάρχουν τεράστιες ανισότητες στις διάφορες ε, περιφέρειες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα δίκτυα, σε ό,τι αφορά και την ταχύτητα, την ψηφιακή ταχύτητα στις διάφορες περιφέρειες. Υπάρχουν επίσης και διαφορετικά επίπεδα γνώσης σε ό,τι αφορά το πώς μπορεί κανείς να συμμετάσχει ενεργά σε αυτήν την ε, ψηφιακή κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να υπάρχει ίση γνώση και ίση συνδεσιμότητα. Και το τρίτο ζήτημα που θέλω να θίξω, όταν ε, μιλάμε για την ψηφιακή κοινωνία και για την ψηφιακή αγορά, συνήθως αναφερόμαστε σε δίκτυα, σε λογισμικά, σε τεχνικά ζητήματα. Η ειδική γνώση των ανθρώπων του πώς να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν όλες αυτές τις έννοιες είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία πώς να μπορεί να χρησιμοποιεί όλες αυτές τις ψηφιακές ευκαιρίες, ούτω ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στην πολιτική ζωή, αλλά και στην, ε, να εξασκήσει την ελευθερία του λόγου. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Τέλος, θέλω να αναφερθώ και στα ζητήματα προστασίας ε, προσωπικών δεδομένων, αλλά και ασφάλεια στη χρήση των διαφόρων κοινωνικών δικτύων και του διαδικτύου, κάτι το οποίο θα πρέπει να αρχίζει να συμβαίνει από πολύ μικρή ηλικία. Τους πολύ νεαρούς μαθητές θα πρέπει να τους εκπαιδεύουμε στο πώς θα μπορούν να είναι ασφαλείς στην ψηφιακή εποχή. Σας ευχαριστώ, λέει ο μιλητή. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρος, συνάδελφε, για την παρέμβαση εκ μέρους των Πρασίνων. Επόμενος ομιλητής στη λίστα μου από την ΚΟΕ, η κυρία Ματίας. Έχετε το λόγο. Η κυρία Ματίας ήταν παρούσα μέχρι πριν λίγο. Η κυρία Τόια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις σχετικά με το θέμα το διαδικαστικό που έθεσε ο Ζωρίνιο έτσι ώστε να αποφύγουμε κάποια στοιχεία σύγχυσης. Γύρω από τις ε, παρατηρήσεις επί της ουσίας άκουσα προσεκτικά ε, τον συνάδελφο που αντικαθιστά τον εισηγητή και θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Καταρχάς, ε, ψηφιακές υπηρεσίες από πλευράς της δημόσιας διοίκησης. Νομίζω ότι αυτή η ψηφιοποίηση θα πρέπει να καλύψει συγκεκριμένα τις ανάγκες των τομέα αυτό, γιατί παρέχονται υπηρεσίες όχι μόνο ενημέρωσης, αλλά γενικότερα υπηρεσίες προς τους πολίτες, και βοηθούν τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν, να ενημερωθούν και ανοίγουν ένα πολύ σημαντικό πεδίο το οποίο μέχρι τώρα τους ήταν κλειστό και δεν μπόρεσε να καλλιεργηθεί ως όφιλε. Δεύτερον, θα ήθελα να διευκρινίσουμε λίγο εδώ την πιθανή διεύρυνση των υπηρεσιών και των δράσεων της ψηφιοποίησης για να βελτιώσουμε την ποιότητα της δημοκρατίας να υπάρξει δηλαδή ήδη από την αρχή των σχολικών προγραμμάτων μία προσπάθεια βελτίωσης των δημοκρατικών κανόνων, να υπάρχει μία συνεχής ενημέρωση, μία κατάρτιση γύρω από τα θέματα αυτά και για αυτούς που ασχολούνται με την τεχνολογία την ψηφιακή, με την κουλτούρα αν θέλετε την ψηφιακή, και γενικότερα με το σύνολο των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Πολλοί πιστεύουν ότι οι διάφορες πλατφόρμες των μέσων ενημέρωσης και τα λοιπά και επικοινωνίας θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο ενημέρωσης για τους πολίτες έτσι ώστε να είναι σε θέση σε τεχνικό επίπεδο να χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά και να γνωρίζουν επί της ουσίας τι σημαίνει η χρήση αυτών των αυτών των δυνατοτήτων συμμετοχής στις ψηφιακές κοινότητες. Όταν μιλάτε για τη σπονδυλική στήλη του συστήματος αυτού, δημιουργείται μία μικρή ε, σύγχυση. Ε, ίσως ε, η κυβερνοασφάλεια, ίσως ε, τα ευφυή e e συστήματα επικοινωνίας, ίσως κάποιες άλλες πλευρές μπορεί να θεωρηθούν από μόνες τους σημαντικές και γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε τους διαχωρισμούς αυτούς και θα πρέπει το σύνολο να διδάσκεται στους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να έχει ζητήσει το λόγο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια παρατήρηση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Φεράρη παρακαλώ έχει το λόγο από την Αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους ε, για τις υποδείξεις και τις ε, απόψεις πολύ εύστοχες ε, και έχουν και μεγάλη σχέση με το περιεχόμενο του σχέδιου δράσης Κομισιόν. Από πλευρά μου θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι ψηφιακέ δεξιότητε δεν είναι σημαντικέ μόνο για τι ε, μελλοντικέ ε, θέσει εργασία ε, και τη ζωή στο μέλλον, αλλά ήδη από σήμερα, γιατί χωρί την τεχνολογία δεν μπορεί κανεί να εργαστεί ούτε να ζήσει σωστά. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν διάφορε ενέργειε προ αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά οι ψηφιακέ ικανότητε εντάσσονται στι βασικέ ικανότητε για τη διαβίου ε, μάθηση. Το σχέδιο δράση βασίζεται κυρίως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εστιάζει και στην ανώτερη βέβαια. Αναγνωρίζουμε όμως τη σημασία της διαβίου μάθησης και της ανάγκης να αποκτηθούν νέες δεξιότητες, να βελτιωθούν ήδη υπάρχουσες, όχι μόνο για τον επαγγελματικό βίο, αλλά και για το βίο εν γέννη, όπως είπα. Ψηφιακές δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές σήμερα για την πολιτική συμμετοχή, τη δημοκρατική συμμετοχή. Επομένως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι Είμαστε πολίτες, αλλά πρέπει να είμαστε και ψηφιακοί πολίτες. Οι ψηφιακές τεχνολογίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη συμμετοχή μας στα δρόμενα, αλλά και στις δημόσιες υπηρεσίες και τις πολιτικές υπηρεσίες. Η εκπαίδευση είναι κλειδί. Δύο ακόμα σχόλια. ψηφιακές δεξιότητες θεωρούμε ότι είναι μια ευρεία δέσμη δεξιότητων που όλοι πρέπει να έχουν σήμερα και σε όλη τη διάρκεια τη ζωής. Υπάρχουν όμως και εξειδικευμένε δεξιότητες στον τομέα τεχνολογιών πληροφοριών επικοινωνίων που πρέπει να αποκτηθούν. Δεν μιλάμε για δεξιότητε που έχουν να κάνουν μόνο με προγραμματιστέ ή ειδικού σε θέματα ψηφιακών τεχνολογιών. Σήμερα το να έχει κανεί ψηφιακέ δεξιότητε υψηλέ δε σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζει σε βάθο ε, ε, πράγματα που μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλού τομεί, όχι μόνο στον τομέα τεχνολογιών πληροφοριών επικοινωνιών. Μπορεί να είναι ψηφιακό καλλιτέχνη, αναλυτή, κάποιο κτλ. Και βέβαια, ψηφιακή εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική για όλα αυτά, διότι δημιουργεί καινοτομία στην εκπαίδευση και πολλά υπουργεία, πολλά κράτη ε, ήδη μετασχηματίζονται και αλλάζουν για να μην μείνουν πίσω και να ακολουθήσουν τους ρυθμούς της σύγχρονης κοινωνίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις παρατηρήσεις σας, κυρία εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνάδελφε Ντέλη, που εκπροσωπείτε τον εισηγητή μας. Ναι. Μάλλον πολλοί εκπροσωπούν πολλούς εδώ, γιατί όλοι ε, κάποιον αντικαθιστούν σήμερα εδώ. Αλλά τέλος πάντων, για να ολοκληρώσω εκ μέρους του κυρίου Ντόιτς, κατά κάποιο τρόπο, Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους, για τα σχόλιά τους. Εκ μέρους του κύριου Ντόιτς λέω ότι φυσικά και θα συνεργαστεί και στο πλαίσιο της διαδικασία ε, κατάθεση τροπολογιών για την επίτευξη συμβιβασμών. Ευχαριστώ. Education, youth, sport, culture, world. Εκπαίδευση, πολιτισμός, ε, αθλητισμός, ε, μπορεί να μην είναι μόνο αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανεί κάτι για του τομεί αυτού και να μπορεί να επηρεάζει τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε, προθεσμία κατάσταση τροπολογιών είναι η 5η Σεπτεμβρίου του 2018. Ψηφίζουμε στις 14. Και πάμε στο επόμενο σημείο που είναι η μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. Θα συζητήσουμε το σχέδιο γνωμοδότηση. Κυρία Μπάρμπαρα Κάπελ είναι η συγγήτριά μας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η μείωση της ποσότητας θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων που έρχονται από, από πλαστικά μιας χρήσης και από ελευτικά εργαλεία που ε, περιλαμβάνουν πλαστική ύλη, συμπληρωματικό μέτρο στο πλαίσιο της στρατηγικής ε, της Ένωσης για τα πλαστικά. Πριν από τις τερινές διακοπές μας ε, έκανε μια πρώτη παρουσία στο σχέδιο γνωμοδότησης η συγκεκριά μας με στόχο να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ταχεία υιοθέτηση αυτής για να έχει και η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή έμβη τον χρόνο που χρειάζεται για να προβεί στις διαπραγματεύσεις πριν το τέλος της θητείας. Δεν έχει δηλαδή απομείνει και πάρα πολύ καιρός. Κυρία Ισηγήτρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε λοιπόν αυτό το σχέδιο πρότασης ε, για μια οδηγία για την πρόληψη και μείωση θαλάσσιας ρήπασης από πλαστικά απορρίμματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν λάβουμε υπόψη τα εκατομμύρια των τόνων πλαστικών απορριμμάτων που ρίχνονται στους ωκεανούς και αποτελούν σημαντική απειλή για τα οικοσυστήματα και τη βιοπικιλότητα, για την ανθρώπινη υγεία, για τον τουρισμό, για την αλία και την ε, ναυσιπλοεία. Είναι ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά Οκτώ από τα 20 σημαντικότερα ε, μολύνοντα κράτη είναι η Κίνα, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Βιετνάμ, ε, αλλά και η ΙΠΑ. Είναι δηλαδή χώρες που δεν ε, ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από το 80% των θαλάσσιων απορριμμάτων προέρχονται από τις 20 αυτές χώρες που δεν είναι από την Ένωση. Και αυτό είναι θετικό τουλάχιστον. Θέλουμε λοιπόν να περιορίσουμε τη θαλάσσια ρηπάνση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε δράση σε επίπεδο G7, G20 ε, της Παγκόσμιας Σύμπραξης κατά των θαλασσίων απορριμμάτων. Δηλαδή είναι μια γενική προσπάθεια αυτή που θα πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το πρώτο. Ε, το δεύτερο είναι ότι θέλουμε ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας ή δυνατόν σε παγκόσμιο επίπεδο ε, για να μειωθούν τα θαλάσσια απορρίμματα και η κυκλική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέλουμε να έχουμε ένα στόχο 50% για την ανακύκλωση μέχρι το 2050 και 55% μέχρι το 2030. Αυτό είναι σίγουρα ένας, μεγάλος, ένας πολύ φιλόδοξος στόχος που είναι όμως ε, δυνατό να επιτευχθεί. Θέλουμε και ε, μείωση ε, σημαντική του 2000, το 2030 σε σχέση με το 2010. Υπάρχουν προτάσεις ε, της Κομισιόν, έχουν δημοσιοποιηθεί, τις συζητούμε σήμερα. ορίζονται δε σε αυτήν την ανακοίνωση τα 10 ελαστικά αντικείμενα μιας χρήσης ε, τα οποία ε, δημιουργούν ε, την μεγαλύτερες ποσότητες τέτοιων πλαστικών όπως είναι περιέκτες, ροφήμων, πλαστικές φιάλες κτλ. Αλλά και στα αλλιευτικά εργαλεία υπάρχουν τέτοια πλαστικά, τα μακροπλαστικά τα οποία δημιουργούν αυτή την ρήπανση. Ε, και θέλουμε να έχουμε μειώσει ε, κατά το ίμιση αυτά τα ε, απορρίμματα. Και υπάρχει και η διάταξη της απαγόρευσης ορισμένων τέτοιων πλαστικών. Εμείς θεωρούμε όμως ότι ένα σημαντικό στοιχείο είναι να δοθούν και κίνητρα για την χρήση αλληλευτικών εργαλείων χωρίς πλαστικό από τους αλληλείς και γενικώ να ε, υπάρχουν ε, μειώσεις ε, της χρήσης. Πιστεύω ότι θα έχουμε έτσι πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση. 11 δις θα εξοικονομηθούν, θα μειωθούν πάρα πολύ οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα με το 2030. Σίγουρα ε, θα υπάρξουν και εξοικονομήσεις για τους καταναλωτές γύρω στα 6,5 δισεκατομμύρια. Η Επιτροπή θεωρεί ότι θα υπάρξουν κάποιο, θα υπάρξει πρόσθετο κόστος για την αλία που είναι γύρω στο 0,16% των εσόδων. Έρχομαι στο τελευταίο μου σχόλιο που είναι η ε, αναλογικότητα και να υπάρχει μία ε, λογική ε, μείωση. Υπάρχουν πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες στήγονται. Για αυτές χρειάζεται χρόνος. Θα πρέπει λοιπόν να ε, είναι σωστές οι προθεσμίες για, τους, ε, για τις υπηρεσίες αυτές. Δεν έχει γίνει ακόμη μελέτη επιπτώσεων, μελέτη αντικτύπου. Πρέπει να υπάρχουν ε, ε, υψηλότερα πρότυπα. Έχουμε την ανάγκη για αβιοαπικοδομήσιμα προϊόντα. Και το τέταρτο, είναι ε, το τέταρτο σχόλιο που έχω να κάνω έχει να κάνει με την έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία σε ό,τι αφορά την στρατηγική για τα πλαστικά. 100 εκατομμύρια θα έχουμε μέχρι το 2020 επιπλέον ο προπολογισμό για την έρευνα και καινοτομία και αυτό είναι θετικό. Να προωθήσουμε βιοαπικοδομήσιμα, βλαβεία, ανακυκλώσιμα προϊόντα και σίγουρα θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας, τουλάχιστον 30.000. Και ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα, το πέμπτο συμπέρασμα, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση ό,τι αφορά ε, αυτή ε, την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών ε, αντικειμένων. Έχω καταθέσει τις σχετικές τροπολογίες και Περιμένω τώρα την ε, ανταλλαγή απόψεων με τους σκιώδεις εισηγητές. Περιμένω τις ε, τροπολογίες και φυσικά και την πρώτη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Εκ μέρους του... Η κυρία, η Σπυράκη εκ μέρους του ΕΛΠ. Ευχαριστούμε πολύ. Πρόεδρε, πρώτα... Is on the Most of the waste does not come from the Ένωσης πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι οποιαδήποτε αποτελεσματική πολιτική θα πρέπει να είναι ένα μείγμα των λεγόμενων τριών E. Πρώτα απ' όλα, engagement, engineering και enforcement. Ενδυνάμωση, α, δημιουργία και δέσμευση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο γνώσης των πολιτών. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά των καταναλωτών για τα συγκεκριμένα προϊόντα, τα πλαστικά μιας χρήσης. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα στην καταπολέμηση της ρήπανσης. είναι ανάγκη να αυξήσουμε την ε, γνώση των πολιτών Κυρίω ξεκινώντα από τα σχολεία και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έχουν λάβει μέρο στην πρωτοβουλία αυτή, να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα α, περήφανη για το βαθμό δέσμευσης. Πρέπει να α, μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε την δημιουργικότητα των διαφόρων επιχειρήσεων. Είναι ανάγκη, ιδίω στον Νότο, να μπορέσουμε να υπογραμμίσουμε τα πλεονεκτήματα που θα μπορέσουν να προκύψουν αν μπορέσουμε να έχουμε καινούριε στρατηγικέ, καινούριε ιδέε. Υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία για να το καταφέρουμε αυτό, όπω για παράδειγμα είναι ο Ορίζον Ευρώπης που επικεντρώνεται στην καινοτομία αλλά και επενδυτικά προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν στην μετάβαση αυτή. Θέλω να σας δώσω ένα νούμερο. Στην Ελλάδα, στην χώρα μου, υπάρχουν περίπου 300 επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου πλαστικά μίας χρήσης και τώρα ψάχνουν για αδιαφορετικού τύπου πλαστικά ανακυκλώσιμα για τις επιχειρήσεις τους. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε 8% ανακυκλώσιμου πλαστικού. Είναι ανάγκη να δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο μας. Γι' αυτό και συμφωνώ με την Επιτροπή που κάνει λόγο για απαγόρευση της χρήσης του πλαστικού. Θέλω να προτείνω συγκεκριμένες ε, διατάξεις για τα νησιά και για τις παράκτιες περιοχές που υποφέρουν περισσότερο από αυτή την μόλυνση. Τέλος, θέλω να πω ότι είναι ανάγκη να αλλάξουμε το καταναλωτικό μοντέλο, αλλά και να προσκαλέσουμε τις τοπικές κοινωνίες για την μείωση της ρήπανσης από τα πλαστικά, αλλά και να προετοιμάσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. αν υπομονώ στη συνεργασία με τους συζητητές σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, για τους φιλελευθέρους. Ρικέ, αντικαθιστά τον Τέλιτσκα. Ζητώ συγγνώμη για τον Πάβελ. Θα διαβάσω όμως την ανακοίνωσή του. Θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή λοιπόν για την προσπάθεια την οποία έκανε, την εισηγήτρια μάλλον. Δυστυχώς ε, η μόλυνση από τα πλαστικά είναι πλέον πάρα πολύ ε, επιβαρυντική για το περιβάλλον. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να ξεπεράσουν το πρόβλημα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει καθυστερήσει και πρέπει να οδηγήσει σε πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές και όχι μόνο στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο γενικά ε, του τοπίου των χώρων μέσα στους οποίους ε, διαβιούμε. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, οι αλλαγές στην νομοθεσία πρόσφατα έχουν αρχίσει να τίθενται σε ισχύ. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες προτάσεων. Η πρώτη αφορά την συλλογή των πλαστικών φιαλών από ποτά αναψυκτικά θα πρέπει να αλλάξει η οδηγία η οποία ε, διέπει τα, συγκεκριμένα προϊόντα. Διερωτώμε λοιπόν αν συνεχιστούν οι συνέπειες της κατάστασης αυτής θα οδηγήσουν επιτέλους στην δημιουργία κέντρων συλλογής των συγκεκριμένων φιαλών. Θα πρέπει να ξεφύγουμε μάλιστα και από την απλή λογική να μιλάμε για πλαστικά μπουκάλια και να μιλήσουμε για κέντρα συλλογής πλαστικών, δηλαδή να μιλήσουμε για την ουσία γενικότερα και όχι για τα επιμέρους μεμονωμένα προϊόντα. Τώρα, θα πρέπει επίσης να υπάρξει σωστή κατανομή των ευθυνών υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις που ορίζουν τον ρόλο και τις ευθύνες των παραγωγών. Δυστυχώς δημιουργείται σύγχυση εδώ. Δεν διευκολύνουμε τους παραγωγούς, δεν δημιουργούμε ένα σαφές πλαίσιο για τις ευθύνες των παραγωγών, για τις παραλήψεις τους κτλ. Ε, θα πρέπει ε, να αναγνωρίσουμε στον συγκεκριμένο τομέα και τις ευθύνες των καταναλωτών. Και τρίτον, τα λεγόμενα soft ε, μέτρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως την έννοια της πρόληψης, η οποία θα αποτρέψει τις στρεβλώσεις στην χρήση ορισμένων τέτοιων προϊόντων νομίζω ότι οι προσπάθειες τις οποίες έχουν κάνει ορισμένες χώρες και κάποια προγράμματα τα οποία ισχύουν σήμερα όπως και κάποιες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ θετικά. Χρειάζεται να γίνουν περισσότερα. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να οδηγήσει σε συμπλήρωση της νομοθετικής αρχιτεκτονικής Ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία την οποία έχουμε για να δράσουμε και οφείλουμε στους εαυτούς μας να μην αποτύχουμε, Πρόεδρε. Thank Thank you, Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας από πλευράς της Γκουε. Ο κύριος Σιλουάγκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα των πλαστικών, δυστυχώς, είναι... έχει δημιουργηθεί πολλά προβλήματα. Και ήταν καιρός ε, που ε, να καταθέσει η Κομισιόν νομοθετική πρόταση για τη θαλάσσια ρήπανση λόγω των πλαστικών. αυτή την πρόταση με τα δέκα αυτά ε, πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης που απαντούν πιο συχνά στη θάλασσα. Νομίζω ότι έχουμε κολληθεί στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν αρκεί. Δεν πρέπει να περιοριστούμε μόνο σε διακοσμητικά μέτρα, αλλά να ενισχύσουμε την πρόταση. Φοβάμαι ότι στο τελευταίο σχέδιο της γνωμοδότησης ε, αποδυναμώνεται η θέση αντίθετα. Ένα παράδειγμα ή μάλλον τρία παραδείγματα για τα οποία νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει κάπως η διατύπωση, να ενισχυθεί. Πρώτον, να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος ε, στην επαναχρησιμοποίηση αυξάνοντα τον αριθμό των, με, των αντικείμενων που θα καλύπτονται και να έχουν ποσοτικοποιημένου στόχου για τη μείωση τη κατανάλωση ε, για του περιέκτε ε, τροφίμων και ποτών. Δεύτερον, να μην υποκατασταθεί η χρήση πλαστικών προϊόντων από τα βιοαπικοδομήσια προϊόντα που πολλές φορές έχουν παρόμοιο αντίκτυπο για το περιβάλλον. Δηλαδή, στόχος εδώ πρέπει να είναι όχι να παραμείνει αυτή η επιβλαβής κουλτούρα του περιέκτη, μέχρι και στις μπανάνες. Στις μπανάνες βάζουμε σε, ε, γύρω από πλαστικά. Ε, αυτή είναι μια κακή πρακτική. Και το άλλο σημαντικό είναι η παραγωγή. Η δευρυμένη ευθύνη παραγωγή. Πρέπει όλοι η παραγωγή να έχουν όλη την ευθύνη ε, όπως ε, και η αρχή ορυπαίνων πληρώνει, κάτι αντίστοιχο. Εμείς θα καταθέσουμε προτάσεις και ελπίζουμε να είναι επικοδομητική η συζήτηση. Ευχαριστώ. Oh, Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε, λέει ο πρόεδρος. Ο Ζωρίνιο, εκ μέρους του των σοσιαλδημοκρατών. Είναι ένας πολύ σημαντικός αυτός ε, τομέας. Ε, είναι, εγώ είμαι και στην Επιτροπή εδώ τακτικό μέλος, έξω και ήθελα να συνεισφέρω και για την έμβη είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πάρα πολύ σημαντικό εν γέννη. Και πρέπει η εκστρατεία μας να είναι πάρα πολύ ισχυρή, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τους ε, συμπολίτες μας, όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Επίσης, πρέπει να δράξουμε αυτή την ευκαιρία για να δώσουμε κίνητρα υπέρ της επαναχρησιμοποίησης ε, των πλαστικών. Θέλουμε να υπάρχει ένα οικονομικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο όποιος ρηπαίνει θα πληρώνει. για να πάψουν να δημιουργούνται πραγματικές ε, ήπειροι από πλαστικά στις θάλασσές μας. Πρέπει να έχουμε μια παγκόσμια στρατηγική για την ανακύκλωση. Πρέπει να είμαστε καινοτόμοι και στον τομέα της αλίας. Πρέπει να βελτιώσουμε την καινοτομία στα αλληλευτικά εργαλεία, να έχουμε επίσης στόχους διαφανείς που μπορούν να μελετηθούν και να αποστικοποιηθούν. και να προωθήσουμε, όπως είπα, και μια ενημερωτική καμπάνια ευαισθητοποίηση, ώστε όλοι μας ε, να ακολουθήσουμε μια διαφορετική ε, συμπεριφορά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε. Έχει ενδιαφέρον να είναι κανείς μέλος και των δύο επιτροπών και της ΕΝΒΗ και της ήτρε και να παρακολουθεί τις συζητήσεις για τα ίδια θέματα και στις δύο επιτροπές. Μου έχει τύχει. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την γνωμοδότησή της, η οποία θα βοηθήσει την συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει σε πολλές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια συζήτηση που θα μας βοηθήσει να τηρήσουμε και το αυστηρό διάγραμμα που έχουμε. Στην παρούσα φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως ακούει ακούει για να κατανοήσει ε, τα κίνητρα και τις, ε, το τι βρίσκεται πίσω από τις προτάσεις. Υπάρχουν όμως κάποιες προκαταρκτικές κρίσεις και για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και για τα σχόλια τα οποία ακούστηκαν πολύ σήμερα. Με ικανοποίηση σημειώνουμε ότι υπάρχει μια ισχυρή στήριξη στην αντιμετώπιση της μόλυνσης ε, της ε, θάλασσας και υπάρχουν προτάσεις ε, διαφοροποιούμενες μεταξύ τους για τα μέσα για να το πετύχουμε. Η σφαιρική καταπολέμηση της μόλυνσης από τις πλαστικές ουσίες δεν είναι κάτι που αφορά μόνο στην Ευρώπη αλλά και την Ασία και στην Ασία και σε άλλες περιοχές του κόσμου και γι' αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε το λεγόμενο global approach έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα πλαστικά και τα λεγόμενα μικροπλαστικά. Είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες οι οποίες ε, βέβαια κυρίως δημιουργούνται στην Ευρώπη, από την Ευρώπη και εις βάρος της Ευρώπης και θα επανέλθω στις προτάσεις του Αντιπροέδρου Τίμερμανς, ο οποίος είχε πει ότι απαιτείται μια νέου τύπου συνεισφορά στην δημιουργία λύσεων για το συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο έτσι κι αλλιώς εμείς εν δημιουργούμε. Γι' αυτό που ακούσαμε σήμερα, καλό θα είναι να τα δούμε μαζί με τις προτάσεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει μέχρι τώρα εμείς έχουμε ορίσει κάποια προϊόντα, περιορισμένο κατάλογο, τα οποία βρίσκονται σε ακατάλληλους ε, περιέκτες, σε ακατάλληλες συσκευασίες όπως ε, προϊόντα προσωπικής υγιεινής Από τη μία δηλαδή υπάρχει η αντίληψη της μίας πρότασης που θα καλύπτει όλα τα προϊόντα και από την άλλη κάτι το οποίο είναι πιο πρακτικό, μία πρόταση για κάθε προϊόν. Συνεπώς λοιπόν είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει τους εναρμονισμένους κανόνες μέσα από μια κατεξουσιοδότηση ε, πράξη. Τώρα για το περιεχόμενο σε πλαστικά των προϊόντων είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ανησυχίες γιατί ορισμένα προϊόντα ακριβώς το ότι αποτελούνται από πλαστικά καθορίζει την καταλληλότητα ή ακαταλληλότητα της απόσυρσής τους. Εμείς δεν είμαστε εναντίον των πλαστικών γενικά, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να ορίσουμε κάποιους τομείς τους οποίους τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να αποσύρονται. Νομίζω ότι με τις προτάσεις τις οποίες κάνουμε, ιδιαίτερα στο άρθρο 15, στοχεύουμε στη μείωση της παραγωγής των προϊόντων αυτών και στα πλαίσια της παρακολούθησης και της στρατηγικής ευρύτερα για τα πλαστικά αντιμετωπίζοντας κάποιες από τις προτάσεις, οι μελέτες επιπτώσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα δείχνουν ότι οι εκστρατείες ενημέρωσης και συνειδητοποίησης είναι ε, συνοδευτικά μέτρα, όχι όμως κάτι το οποίο από μόνο του θα δώσει λύση. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας, λέει ο Πρόεδρος, η συγγήτρια έχει το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους σκιώδες εισηγητές για τις πάρα πολύ αξιόλογες παρεμβάσεις τους και βλέπω ότι υπάρχει συμφωνία ως προς το ότι είναι ένα θέμα παγκόσμιο, πολύ σημαντικό. Βιομηχανία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν απαραίτητο, τον απαραίτητο χρόνο στη θέση τους για να αναζητήσουν εναλλακτικές Σίγουρα είναι απαραίτητα τα πρότυπα, σίγουρα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά, ε, και παγκόσμιο, αλλά τέλο πάντων τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό, αλλά χρειάζεται χρόνο για την εφαρμογή αυτών των προτύπων. Ξέρουμε ε, πόσο σημαντική είναι και η πλαστική βιομηχανία. Ε, και πάρα πολύ σημαντικό είναι να γίνει ε, μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης ε, υπέρ της ανακύκλωσης κατά της αυξημένης χρήσης των πλαστικών και στο πλαίσιο του πακέτου για τη γενική οικονομία ε, και για τα μικροπλαστικά πρέπει να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ε, και βλέπω να υπάρχει συμφωνία με τους κοιοσυγητές. Θα τα δούμε και με τους κοιόδης. Έχουμε ε, σύντομες προθεσμίες. Αύριο λίγη η προθεσμία των καταστροπολογιών και στις 24 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα και επειδή είναι ο χρόνος περιορισμένος, ε, θα πρέπει να υπάρξει ένας δομημένος, ε, μια δομημένη συμβολή και συνεισφορά προς την Καθήλυνα Διευθυντροπή και γι' αυτό ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία του Σκιώδης. Ευχαριστούμε για όλα σας τα σχόλια, αλλά και για το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάσατε. 6 Σεπτεμβρίου, λήξη προθεσμίας για κατάθεση τροπολογιών, λέει ο Πρόεδρος. Και ολοκληρώσαμε και το σημείο 5. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Σε ένα λεπτό ευελπιστώ ότι θα έχουμε όλα μας τα μέλη στην αίθουσα γιατί προς το παρόν δεν είμαστε αρκετοί για να ψηφίσουμε. Good afternoon. Καλησπέρα, συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Κάποιοι από εσά γνωρίζουν ήδη ότι την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, είχαμε μια κοινή συνέλευση με την Επιτροπή Μεταφορών, μια μισή ώρας. Ήταν η πρώτη συνάντηση μετά τις διακοπές. Αυτή είναι η πρώτη συνάντηση της δικής μας Επιτροπής, της Ήτρε. Πιστεύω ότι χαίρεστε που επιστρέψατε. Επιτρέψτε μου να πω, έχουμε σχεδόν έξι μήνες δραστηριοτήτων μπροστά μας. Και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε τον επόμενο μισό χρόνο ως Επιτροπή Ήτρε, γιατί είμαστε υπερβολικά, έχουμε ένα υπερβολικά βαρύ πρόγραμμα, η επιλογή σας τέσσερα χρόνια πριν ήταν άριστοι να είστε μέλη αυτής εδώ της Επιτροπής. Έχουμε 18 νομοθετικούς φακέλους διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο, 18. Επιτρέψτε μου να πω, δύο τριμερείς διαλόγους για κάθε νομοθετική πρόταση. Αυτό τι σημαίνει, 36 διαπραγματεύσεις. Δύο συναντήσεις για κάθε πρόταση. Και για κάποιους φακέλους μπορεί να χρειαστούν τέσσερις συναντήσεις για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το ψηφιακό θεματολόγιο ή ό,τι αφορά προγράμματα πλαίσια. πολύ δουλειά μπροστά μας λοιπόν. Έχουμε 11 νομοθετικές προτάσεις υπό προετοιμασία στα πλαίσια της Επιτροπής, δεν είναι ακόμη έτοιμες. Επτά βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και 11 είναι σε φάση προετοιμασίας. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές και ενώ βλέπω ικανοποίηση στα πρόσωπά σας, χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Πρέπει να ξεκινήσουμε τη σκληρή μας δουλειά με την ψηφοφορία. Ας κάνουμε μια δοκιμή. Άρχεται η ψηφοφορία. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Έχουμε... Έχουμε την ψηφοφορία. Έχουμε τέσσερις προτάσεις. Υποψηφοφορία. Δύο ψήφοι έχουν να κάνουν με την α, ψηφιακή αξιολόγηση και την COP24, ψηφοφορίες οι οποίες έχουν αναβληθεί από τη συνάντηση του Ιουλίου. Θέλω να σας ενημερώσω όλους ότι το πρώτο κομμάτι της αξιολόγησης των τεχνολογιών της υγείας ξεκίνησε την 10η Ιουλίου και η ψηφοφορία θα ξεκινήσει από την τροπολογία 133. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή από την τροπολογία 133. Οι προηγούμενες τροπολογίες έχουν ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. Οι εισηγητέ έχουν ενημερωθεί για, την, ε, για το μερικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Αυτές είναι πολύ σημαντικές πληροφορίες. Από άποψη διαδικαστική λοιπόν είμαστε σε πολύ καλή φάση. Ξεκινάμε με το σημείο 6. Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας. Τροπολογία 133. Υπέρ. Εναντίον. Αποχές. Υιοθετείτε. 134. Υιοθετείτε. Συμβιβασμός 25. Ηλεκτρονική ψήφο γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρη πλειοψηφία. η ψηφοφορία. Γίνεται αποδεκτός. 20 υπέρ. Εναντίον. Να το ελέγξουμε και πάλι ηλεκτρονικά. Ολοκληρώνεται. Απορρίπτεται. Είναι δύσκολο να καταμετρήσουμε. Λέει ο πρόεδρος. 136 υπέρ. Αποδεκτή. 136 αποδεκτή. 138 αποδεκτή. 139 απορρίπτεται. 140 αποδεκτή, συμβιβασμός 26, αποδεκτός, 142, να το ελέγξουμε, τροπολογία 142. Γίνεται αποδεκτή η τροπολογία. 143. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 27, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συμβιβασμός 27. Γίνεται αποδεκτός. 146 τροπολογία. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 146. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 28. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συμβιβασμός 28. Απορρίπτεται. Τροπολογία 147. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 147. Γίνεται αποδεκτή. 23. 148. Απορρίπτεται. 149. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 1. Αποδεκτός. 27 αποδεκτός. Συμβιβασμός 2. Αποδεκτός. 29 τροπολογία. Αποδεκτή. Συμβιβασμός 3. Αποδεκτός. Τροπολογία 32. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρόεδρε, γιατί δεν έγινε ψηφοφορία για την τροπολογία 1... Η τροπολογία 1 λέει ο πρόεδρος καλύπτεται από τον συμβιβασμό 3. Δεν πιστεύω ότι καλύπτεται. Τουλάχιστον στη λίστα που έχω εγώ στα χέρια μου. Υπάρχει πρόταση να ψηφίσουμε για την τροπολογία 1 λοιπόν. Εντάξει, λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 32. Υπέρ. Γίνεται αποδεκτή. Τροπολογία 33. Αποδεκτή. 2. Νούμερο 2. Απορρίπτεται. Τροπολογία 34. Αποδεκτή. Συμβιβασμός 4. Αποδεκτός. 3. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 5. Αποδεκτός. Τροπολογία 40. ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 40. Απορρίπτεται. Τροπολογία 41. Και πάλι ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 41. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42. Ηλεκτρονική ψηφοφορία και πάλι. Γίνεται αποδεκτή. Συμβιβασμός 6. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ολοκληρώθηκε. Γίνεται αποδεκτός. Ο συμβιβασμός 6. Συμβιβασμός 7. Αποδεκτός. Τροπολογία 50. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Απορρίπτεται η τροπολογία 50. Συμβιβασμός 8, ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Γίνεται αποδεκτός. Τροπολογία 52. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 52. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 9. Αποδεκτός. Τροπολογία 24. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Θεωρούνται ε, για το πόσο θα γίνουν αποδεκτές οι τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Ολοκληρώθηκε. Αποδεκτές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και τώρα... Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο όπως και πριν τις διακοπές. Συγχαρητήρια. Επόμενη ψηφοφορία. Πάμε κατευθείαν. Έχουμε μία ψηφοφορία ηλεκτρονική. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Η πλειοψηφία υπέρ. Θα στείλουμε τις γνωμοδοτήσεις μας πέρα από το τυπικό της διαδικασίας, αλλά με πλήρη ε, συμφωνία μεταξύ των συντονιστών, ότι χρειάζεται μια τέτοιου τύπου διαδικασία, αν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι πριν την ψηφοφορία της ΕΝΒΗ, που είναι πριν την προηγούμενη εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, με συγχωρείτε, ούτως ώστε να έχουμε πιο βραχείς διαδικασίε. Όπως βλέπετε όμως, η πλειοψηφία είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο λοιπόν. Και αυτά που θα στείλουμε στην Επιτροπή ΕΜΒΗ είναι πολύ σημαντικά πριν την COP24. Από την ε, οπτική γωνία του τομέα της ενέργειας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της βιομηχανίας, πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να στείλουμε τις γνωμοδοτήσεις μας στους συναδέλφους στην Επιτροπή ΕΝΒΗ. Περνάμε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης, ο Άλντο Πατριτσέλο για την συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το βασίλειο του Μαρόκο. Θυμόμαστε και τη συζητήση μας πάνω στην υπόθεση της πρίμα, της εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και του βασίλειου του Μαρόκο. Τροπολογία νούμερο 1. Υπέρ, εναντίον, αποχές απορρίπτεται. Καθολική ηλεκτρονική ψηφοφορία για το νομοθετικό σχέδιο. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Με πλειοψηφία συγχαρητήρια γίνεται αποδεκτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελείωσε η διαδικασία της ψηφοφορίας, λέει ο Πρόεδρος. Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους που θέλουν να παραμείνουν μαζί μας να παραμείνουν και οι υπόλοιποι να αποχωρήσουν. <laughs> Okay. Well, it was quite clear announcement for myself. Τα είπα πολύ ωραία, έτσι δεν είναι. Ε? Great. Μάλιστα, πολύ ωραία. Να περάσουμε στο σημείο 9 παρακαλώ, της ημερησίας διάταξης θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027. Προσεχές πολιετές νοσονομικό πλαίσιο. Το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη είναι φάκελο στο πλαίσιο του Πολιετές νοσονομικού πλαίσιου. Βασίζεται στην υπολογιστική ψηλών επιδόσεων αυτή την πρωτοβουλία 9 δις λίγο πολύ ευρώ. Είναι ο συνολικός προπολογισμό για τη στήριξη της ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, έρευνας, διατήρηση του ρυθμού που έχουμε σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το γνωρίζουμε. Η συγγετριά μας είναι η κυρία Αγγέλη Καμλίναρ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο. Θέλω να καλωσορίσω τους συναδέλφους που ελπίζω να γύρισαν ανανεωμένοι από τις διακοπές τους. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να σας παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσης για το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη σήμερα. Κάρπο μιας πολύ εντατική δουλειάς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εφόσον έπρεπε να έχουμε έτοιμη την θέση του Κοινοβουλίου και ελπίζουμε και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου πριν το τέλος της θητείας. Φιλόδοξο στόχο. Ελπίζω να επιτευχθεί. Η πρόταση αυτή αφορά το πρώτο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα της Ψηφιακή Ευρώπη. Είναι ένα πρώτο βήμα προς την ενίσχυση και τη βελτίωση της ηγετική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κάλυψη του επενδυτικού κενού που αντιμετωπίζουν στον τομέα αυτό και που επηρεάζει και το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη καινοτόνων ψηφιακών λύσεων και για να αντιμετωπιστεί και η έλλειψη που έχουμε στο επίπεδο αυτό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δηλαδή. Πρέπει να τονίσουμε σε σχέση και με τι προτάσει τη Κομισιόν ότι ο προπολογισμό, το είπατε και εσεί, κύριε Πρόεδρε, ανέρχεται σε 1,2 δι. Αυτό προτείνει η Κομισιόν. Για μα είναι το ελάχιστο ποσό, αν θέλουμε η υλοποίηση του προγράμματο να στεφθεί με επιτυχία. Φαίνεται δυνητικά όμω περιορισμένο αυτό ο προπολογισμό για την επίτευξη των ε, φιλόδοξων στόχων και την αντιμετώπιση προκλήσεων που μπορεί να μην μπορούμε σήμερα να προβλέψουμε. Στο επόμενο πολιετέ θα συνεπάρχει αυτό το πρόγραμμα με άλλε δράσει αφαιρωμένε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Έχοντα υπόψη δε και του μεσομικού περιορισμού από το πολιετέ μεσομικό πλαίσιο, πάρα πολύ σημαντικό, η ψηφιακή Ευρώπη εφαρμοζόμενη σωστά να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματά της και να μην υπάρχει άλλη επικάλυψη με άλλα προγράμματα, αλλά ανάπτυξη ενεργειών. Η βέλτιστη διαχείριση λοιπόν της χρηματοδότησης ε, θα γίνεται με άμεση διαχείριση από την Κομισιόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπήρξε διάλογος με την Κομισιόν μετά από αυτό το διάλογο. Και έχοντας υπόψη μας πόσο ιδιαίτερος είναι κάθε στόχος, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση ανά στόχο. Και αυτό θα γίνει ως εξής. Πρώτος στόχος για την υπολογιστική ψηλών επιδόσεων. Διαχείριση θα γίνει από την νεοσταθή σύμπραξη, κοινοπραξία. Δεύτερος στόχος, για την τεχνητή νοημοσύνη. Διαχείριση από την Κομισιόν. Τρίτος στόχος, κυβερνοασφάλεια. Διαχείριση κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου με βάση το νέο κανονισμό που θα δημοσιοποιηθεί από την Κομισιόν σύντομα, ελπίζουμε. Τέταρτο, για ψηφιακέ δεξιότητε προηγμένε. Και πέμπτο στόχο, ανάπτυξη των πρώτων τριών στόχων. Εδώ η διαχείριση θα γίνεται από του νέου κόμβου Ευρωπαϊκής Καινοτομία. ψηφιακής καινοτομίας. Πρώτη πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, όπω είπαμε, ειδικά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Δύο είναι τα βασικά, οι βασικοί άξονες. Όπου αποδείχθηκαν ανεπαρκείς οι μεμονωμένες δράσεις των κρατομήλων. Πρώτος άξονας, να έχουμε αυτονομία από στρατηγικής πλευράς ό,τι αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες. Επειδή υπάρχουν πολλέ επιλέξιμε δραστηριότητε, δεν θέλουμε να υπάρξει διασπορά. Άρα θέλουμε να υπάρχει νομιλευτικό έλεγχο και σε ό,τι αφορά το κατάρτιση των προγραμμάτων εργασία. Επίση, πέντε είναι οι στόχοι τη Κομισιόν. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με μία μόνη προσέγγιση. Ιδίω αν θεωρήσουμε ότι κάποιοι στόχοι θέλουν να δημιουργήσουν ευρωπαϊκέ δυνατότητε κυρίω, όπω είναι η υπολογιστική υψηλών Αλλά υπάρχουν στόχοι που έχουν να κάνουν με πολύ λεπτού ευαίσθητου τομεί, όπω είναι η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, ή η κυβερνοασφάλεια. Άρα, έχουμε αντιμετωπίσει με το εξή λεπτό ζήτημα στο Κοινοβούλιο. Πώ θα υπάρξει στρατηγική αυτονομία και ελευθερία δράση σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα, μεγάλο προβληματισμό για το πώ μπορούμε να υλοποιήσουμε και να ε, πραγματώσουμε του τρει βασικού στόχου, αλλά και το βασικό στόχο του προγράμματο. Για να απαντήσω το ερώτημα, επικεντρώθηκα στην επιλεξιμότητα των οντοτήτων, αλλά άφησα ανοιχτό και το ενδεχόμενο συνεργασιών με συνδεδεμένες τρίτες χώρες. Ο στόχος μου δεν είναι να υπάρξει από προεπιλογή αποκλεισμό αυτών, αλλά επειδή είναι πολύ διαφορετική μεταξύ τους οι στόχοι, πρέπει να το συζητήσουμε αυτό και να δούμε πώς προσεγγίζουμε το θέμα της εφαρμογής. Εξατομικευμένα και όχι γενικευμένα για όλους το ίδιο τους στόχους. Στόχος μου είναι να περικεράσουμε τα προβλήματα με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Δεύτερη ο σάξονας, δεύτερη διάσταση. Θέλουμε να προωθήσουμε τα ωφέλη της έρευνας καινοτομίας ανάπτυξης. Την τεχνολογία εχμής που θέλουμε να έχουν δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτό το δίκτυο των κόμβων ψηφικής καινοτομία που θα καλύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επικράτεια για να αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων περιβαλλόντων. Ένα κόμβο πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον σε κάθε περιφέρεια. Είναι πρόκληση αυτό, αλλά πρέπει να το επιτύχουμε. Τέλο. Ένα άλλο νοστιό Για να αντιμετωπίσουμε την ιδιαιτερότητα του στόχου τη τεχνητή νοημοσύνη. Ειδική αναφορά στην ηθική συμμόρφωση, δεντολογική συμμόρφωση με βάση και άλλες προτάσεις στο πλαίσιο του πολιετούς μεσορικού πλαισίου. Αυτά περιμένω τις προτάσεις σας και προσβλέπω και σε μια επικοδομητική συζήτηση με τους κοιόδες και τους υπόλοιπους συζητητές. Ah, σας ευχαριστούμε πολύ για τον μακροσκελέστατο λόγο. Δεν σας είχα βάλει χρονικό περιορισμό επειδή ελπίζω ότι έχουμε αρκετό χρόνο. Κύριε Ρούμπικ, εκ μέρους του... του ΕΛΚ. Ευχαριστώ την Δεκαστήγιο, ε, αντικαθιστώ την Δεκαστήγιο Είναι ένα θέμα το οποίο έθεσε με σωστό τρόπο νομίζω η συνάδελφος Μλίνα. Γνωρίζουμε ότι ο προϋπολογισμός τον οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο ελάχιστος δυνατός και εμείς προσπαθούμε να αυξήσουμε πάντα ε, τον προϋπολογισμό των προγραμμάτων αυτών. βασικός στόχος ε, της ε, δομής του προϋπολογισμού και εδώ συμφωνούμε με την εισηγήτρια πρέπει να υπάρξουν αλλαγές σε σχέση και με τις πιθανότητες συμμετοχής των τρίτων χωρών ιδιαίτερα χωρών από την ε, Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. και άλλες τρίτες χώρες. Λοιπόν, θα πρέπει κατά περίπτωση να βλέπουμε τις περιπτώσεις αυτές και γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε κάποιες επιμέρους τροπολογίες έτσι ώστε να παραμείνει φυσικά το πρόγραμμα αυτό ε, ευρωπαϊκό αλλά να ανοίξει και προς τα έξω. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και όλους όσους πήραν μέρος στην επεξεργασία αυτής της πρότασης. Κύριε Ζωρίνιο, έχουμε καλά αποτελέσματα. Είναι η τρίτη συζήτηση που κάνουμε σήμερα το απόγευμα και εκπροσωπείτε για τρίτη φορά τους σοσιαλιστές, αλλά αυτή τη φορά μάλλον εκπροσωπείτε τον εαυτό σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω πάρει το λόγο και ε, σε προσωπικό επίπεδο. Για πολιτικούς λόγους το κόμμα μου δεν έχει εκφραστεί σε κάποιες τομείς. Ε, συμφωνώ πάντως με τις περισσότερες από τις προτάσεις της ηγήτριας, οι οποίες θα βελτιώσουν τον πρόγραμμα και θα μας δώσουν την δυνατότητα να συνεχίσουμε τις εργασίες μας ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε ψηφιακή οικονομία και τις ε, πιθανές κοινωνικές ε, αλλαγές τις οποίες θα επιφέρει. Νομίζω ότι το κείμενο έχει ήδη βελτιωθεί Πρέπει να σημειώσουμε λοιπόν την βελτίωση αυτή και σε σχέση με το δεοντολογικό του κομμάτι και υπάρχει επίσης και το θέμα των λεπτομερών προγραμμάτων εργασίας που ε, δημιουργούνται και μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα ένα πρόγραμμα το οποίο από πλευράς τεχνικής όμως δεν είναι ιδιαίτερα θα έλεγα πυκνό. Συνεπώς όχι μόνο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την οικονομική πρίκα του προγράμματος αυτού, αλλά να προσπαθήσουμε να προγραμματίσουμε και για το μέλλον έτσι ώστε να δώσουμε δυνατότητες σύγκλησης των οικονομιών των κρατών μελών, να βελτιώσουμε την οικονομία της Ευρώπης στο σύνολό της και κυρίως να παρέχουμε τις απαιτούμενες υπηρεσίες στους πολίτες. Αυτές λοιπόν είναι οι κατευθυντήριες γραμμές ε, για την αξιολόγηση των τροπολογιών. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στην διάθεσή μας, το χρονοδιάγραμμα είναι αρκετά αυστηρό. Σχετικά με την ανταγωνιστικότητα απαιτείται να υπάρξουν σωστές εταιρικές σχέσεις, να υπάρξει βελτίωση και ισορροπημένη αν θέλετε, δυνατότητα πρόσβασης στις χρηματοδοτήσεις. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συνδεθεί και με το ευρύτερο πρόγραμμα Horizon uh, Europe. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ε, ικανοί να γνωρίζουν ποια είναι η στρατηγική την οποία ακολουθούμε ε, και θα πρέπει όλα τα στοιχεία να είναι διαθέσιμα και να επιτρέψουμε στους πολίτες να είναι ενήμεροι. Θα πρέπει να υπάρξει και με τα επιμέρους προγράμματα συντονισμός καλύτερος με τα ταμεία συνοχής με πιο ισορροπημένο τρόπο, να βελτιώσουμε την διαλειτουργικότητα των προγραμμάτων να χρησιμοποιήσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τους περιορισμένους πόρους της Ένωσης, να βελτιώσουμε την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθεί στις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις. Αυτό αφορά όλους τους πολίτες, το σύνολο της οικονομίας και το σύνολο των υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν θα είναι όλοι πιο σωστά καταρτισμένοι και θα λειτουργούν με μεγαλύτερη ασφάλεια χωρίς ε, να γενικολογούμε. Όπως είπα το χρονοδιάγραμμα είναι ιδιαίτερος αυστηρό. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στην διάθεσή μας, Εγώ προσωπικά θα κάνω ό,τι μπορώ έτσι ώστε η ευκαιρία αυτή να δώσει καρπούς. Σας ευχαριστώ. κύριος Φόξ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Η δική μου ομάδα έχει αρκετές ανησυχίες για την πρόταση αυτή. Η ψηφιοποίηση, την προσαρμογή στα νέα μοντέλα εργασίας, ιδίως σε ό,τι αφορά την δημόσια διοίκηση. Βλέπουμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες αυτές. Οι καταναλωτές θα έχουν περισσότερα προϊόντα και καλύτερες επιλογές. Για παράδειγμα, να βοηθήσουμε τους μικρούς επιχειρηματίες να έχουν online υπηρεσίες είναι κάτι το οποίο θα αποβεί εποφελές για τους καταναλωτές. Το βασικό ζήτημα εδώ είναι η εμπιστοσύνη για την ψηφιακή μετάβαση και την κυβερνοασφάλεια. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ζητήσω περισσότερες πληροφορίες από την Κομισιόν σε ό,τι αφορά τον τέταρτο κανονισμό για την κυβερνοασφάλεια. Είναι κάτι θεμελιώδες. Το ζήτημα των δεδομένων είναι εξίσου σημαντικό για το μέλλον της ψηφιακής ε, οικονομίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ό,τι αφορά την αρχή τώρα των ανοιχτών δεδομένων, είναι κάτι το οποίο η ομάδα μου στηρίζει. Καλωσορίζουμε τις προτάσεις ε, των εισηγητών για αυτούς τους κόμβους, αλλά και τα ζητήματα που αφορούν την ε, ηθική είναι ανάγκη να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στην ιδιαίτερη φύση της ψηφιακής Ευρώπης, αλλά και για τις νεόφυτες επιχειρήσεις ακόμη περισσότερο. Διαφωνούμε όμως με τον εισηγητή, διότι πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει στρατηγικό στόχος στην πρόταση αυτήν. Δεν από στρατηγική άποψη, δεν συνάδει με κάποιες ε, στρατηγικές ανησυχίες που σε τελική ανάλυση θα πρέπει να προκύψουν περιορίζοντας συγκεκριμένα κομμάτια του προγράμματος αυτού σε ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες ασφαλείας και συγκεκριμένα σε ιδιαίτερους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης θεωρούμε ότι ίσως και να υπάρχουν κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια. Δεν βλέπουμε τον κίνδυνο στην επιπλέον κατάρτιση των εργαζομένων, ψηφιακή κατάρτιση ή στην εγκατάσταση προγραμμάτων αντιβάρους. Πιστεύουμε ότι η ψηφιακή Ευρώπη θα μπορούσε να είναι ένα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα και ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να εργαστούμε από κοινού και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε λέει ο Πρόεδρος. Ηθικά ζητήματα είναι πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά την ψηφιακή Ευρώπη. Ο επόμενος ομιλητής Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαστε πεπισμένοι πως η ψηφιοποίηση, το βιομηχανία 4.0 και άλλες αναφορές στις ψηφιακές αυτές αλλαγέ στο ψηφιακό μετασχηματισμό πρέπει να είναι πηγές ευκαιρία. Αλλά πρέπει να υπάρχει δημόσια πολιτική διαχείριση αυτών των αλλαγών που θα ωφελεί την πλειονότητα των συμπολιτών μας. Η επιχειρηματική λογική που εφαρμόζεται στην ψηφοποίηση λέει ότι όποιοι ε, προσαρμόζονται επιβιώνουν και όσοι αντιστέκονται πεθαίνουν. Αυτό δεν μπορεί να είναι η κοινωνική δημοκρατική λογική ε, των κρατών δικαίου. Υπάρχει συνένεση ως προς το ότι το λιγότερο σημαντικό στην ψηφιοποίηση είναι τα τεχνολογικά. Ε, πολύ πιο αποφασιστικές είναι οι πτυχές ε, της ε, οργανωτικής κοινωνικής δομής και τάξης. Αυτό είναι και το αντικείμενο της πρώτης μου παρέμβασης. Οι ανησυχίες μας εστιάζουν στο ότι θέλουμε να αποφύγουμε η ψηφιοποίηση να διχάσει ακόμη περισσότερο την κοινωνία. Να έχουμε από τη μία τους λίγους νικητές και από την άλλη τους πολλούς ιτημένους και δεν θέλουμε να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανισότητα στην ανακατανομή του πλούτου. Αυτό μα το έχει υποδείξει και η Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Επίση, η διάσταση του φύλου πρέπει να εφαρμόζεται σε όλε τι πολιτικέ. Να είναι κινητήρε, να είναι μοχλό για την ισότητα ανδρών και γυναικών και να καταπολεμάται έτσι το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Επίση, υπάρχει γενεακό χάσμα σε ό,τι αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Υπάρχουν όλο και μεγαλύτερε διαφορέ επίση μεταξύ περιφερειών σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρουν αυτέ οι τεχνολογίε. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια αξιολόγηση της κοινωνικής, ε, των κοινωνικών ε, επιπτώσεων αυτών των κανόνων που επηρεάζουν του εργαζομένου ε, και τον κόσμο τη εργασία εν γέννη. Θα πρέπει λοιπόν να συμμετέχουν κοινωνικοί εταίροι και στι αποφάσει που θα λαμβάνονται. Θεωρούμε σημαντικό να υπάρχουν στοιχεία που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Οι ψηφιακέ ε, υπηρεσίε θα πρέπει να είναι προσβάσιμε, ε, να παρέχονται σε όλου και οι δημόσιε διοικήσει θα πρέπει να παρέχουν στου πολίτε και στου εργαζομένου την απαιτούμενη βοήθεια. Τέλο, οι προτάσει που ε, αναφέρονται στο πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη μπορούν να είναι ένα μεγάλο εργαλείο υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπληρωθούν με κανόνες που θα πηγαίνουν στην κατεύθυνση της συμπερίληψης όλων, δηλαδή να υπάρχει πρόσβαση, να υπάρχει Μείωση των αυξανόμενων ανισοτήτων και διαφορών. Το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, πάντως φαίνεται να είναι κατακαιρματισμένο σε διαφορετικές πρωτοβουλίες που μας δυσκολεύουν να έχουμε μια συνολική θεώρηση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή ποια θα είναι η πραγματική επίπτωση των προτάσεων. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την δυνατότητα που προσφέρει αυτό το πρόγραμμα, αλλά να σκεφτούμε πολύ σωστά τι προτάσεις πρέπει να εφαρμόσουμε και τι επιπτώσεις θα έχουν αυτές για όλη την κοινωνία. Ευχαριστώ. Thank you, madam, for your Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε τον εισηγητή. Θέλω να εφιστήσω την προσοχή σας σε ένα σημείο που δεν θεωρώ ότι το έχει λάβει ε, υπόψη της η Κομισιόν όσο θα έπρεπε. Μιλάω για την ανάπτυξη Τη τεχνητή νοημοσύνης. Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία στην οποία δεν έχουμε δράσει όσο γρήγορα θα έπρεπε. Ο προπολογισμό ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη θεωρώ ότι δεν είναι όσο θα έπρεπε να είναι για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην ευκαιρία αυτή. Είναι ανάγκη να επενδύσουμε παραπάνω στην ε, οικονομία της γνώσης αλλά και για την μελλοντική αυτή εξέλιξη στον τομέα της έρευνας. Ε, σε αυτήν την έκθεση πρέπει να δώσουμε σημασία στην κεντρική διάσταση της ε, τεχνητής νοημοσύνης, κάτι το οποίο μπορεί να αποβεί εποφελές για όλους τους Ευρωπαίους. Θέλω να σας προειδοποιήσω και για την διαδικασία της κανονικοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το φόρουμ που εργάζεται στο τεχνικό κομμάτι της, του τομέα αυτού α, κυρίως δραστηριοποιείται στην Αμερική ή στην Κίνα. Ο τρόπος χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης ε, είναι κάτι το οποίο μπορεί και να περιθωριοποιήσει την Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό ε, πήρα το λόγο γιατί ήθελα να ευαισθήσω την προσοχή σας στο σημείο αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, για τα σχόλιά σας. Η Γενική Διεύθυνση Connect, ο κύριος Βέζα Τέραμπ, εκπροσωπεί την Γενική Διεύθυνση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Έχει προχωρήσει και με μεγάλη ταχύτητα και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση με τους στόχους που έχουμε για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό. Αυτό που είναι ακόμα πιο σημαντικό βέβαια είναι το περιεχόμενο της έκθεσης και εδώ υποστηρίζουμε την στήριξη την οποία παρέχει ο εισηγητής στην πρότασή μας Έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στην Ευρώπη έτσι ώστε να παρέχονται οι απαιτούμενες ψηφιακές δυνατότητες και για τον δημόσιο τομέα και για τις επιχειρήσεις να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιούν σωστά και να ωφελούν τους ε, ε, πολίτες, τους επιστήμονες, τους φοιτητές κτλ. Κάποιες ε, προκαταρκτικές τώρα παρατηρήσεις για τα σχόλια τα οποία προηγήθηκαν. Είναι θετικό για μας που θεωρεί ότι η πρότασή μας είναι η ελάχιστη σε δημοσιονομικό επίπεδο έτσι ώστε να πετύχουμε τις, ε, να αναπτύξουμε τις δυνατότητες αυτές και να δούμε πώς στα πλαίσια του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου θα υπάρξει κατανομή των χρημάτων έτσι ώστε να μην μείνουμε στο ελάχιστο δυνατό το οποίο παρέχεται στην παρούσα φάση. για την πρόταση του εισηγητή τώρα. να υποδειχθεί ήδη στην πρόταση κανονισμού ποια θα είναι τα σώματα τα υπεύθυνα για την εφαρμογή των διαφορετικών στόχων. Αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί ακόμα. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς και τι γίνεται με ε, την πρόταση μελέτης επιπτώσεων η οποία συνοδεύει την πρόταση και να δούμε πώς θα δώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στην πρόταση ανάλογα με την εξέλιξη των δράσεων τα επόμενα χρόνια. Αλλά είναι σαφές ότι θα εμείνουμε στους βασικούς στόχους τους οποίους έχουμε θέσει τώρα. Τα λεγόμενα innovation hubs, τα κέντρα καινοτομίας. Ε, πρέπει να καταστήσουμε διαθέσιμα τα μέσα αυτά και για τους οικονομικούς εταίρους και για το σύνολο των εμπλεκομένων σε διάφορα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρέπει να υπάρξει δηλαδή μια σωστή κατανομή ε, των δυνατοτήτων αυτών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι αυτά τα innovation hubs θα πρέπει να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό δίκτυο έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες οι εμπειρίες και η ε, εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει ε, στο σύνολο των ε, εμπλεκομένων πολιτών και των επιχειρήσεων ε, στα πλαίσια της διασύνδεσής τους. Τώρα για τις υπόλοιπες προτάσεις, στην παρούσα φάση απλά θα ήθελα να πω ότι λαμβάνω υπόψη τις προτάσεις οι οποίες γίνονται θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις τρίτες χώρες και με ποιες δυνατότητες θα μπορούν οι χώρες αυτές να συμμετέχουν. Η συζήτηση η οποία γίνεται είναι αν θέλουμε ήδη να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά στην πρόταση είναι κάτι για το οποίο θα επιφυλαχθούμε σε ιστερότερη φάση να διατυπώσουμε. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα ήθελα να θέσω έγινε μία πρόταση, η τελευταία πρόταση για την τεχνητή νοημοσύνη. Είπατε ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο ποσό. Νομίζω ότι θα πρέπει να ειδωθεί το πρόγραμμα στο σύνολό του. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε βέβαιοι και να ορίσουμε σωστά το σύνολο του προϋπολογισμού και μετά να δούμε ακριβώς ε, ποια ισορροπία θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ανάμεσα στις διαφορετικές ε, μορφές και ανάγκες χρηματοδότησης. είναι κάτι το οποίο θα αναζητηθεί δηλαδή σε έφετο χρόνο. Πάντως γενικά σας ευχαριστώ για τις προτάσεις σας. Πέραν αυτού όμως, εμείς θα συνεχίσουμε τις επαφές έτσι ώστε να βρούμε κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία έχετε μέχρι τώρα διατυπώσει. Σας ευχαριστώ και εγώ για τις παρατηρήσεις σας. τελικές παρατηρήσεις στον εισηγητή μας, στην εισηγήτρια. Μπορεί να μιλάει όσο θέλει, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Τα ΕΠΑ και στην αρχή βέβαια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τους κοιόδης από τις άλλες πολιτικές ομάδες για τη στήριξη συνολικά και για την ε, αφοσίωση τους στο αυτό το πρόγραμμα. Θεωρούμε ότι είναι ένα καλό πρόγραμμα όλοι. Έτσι φαίνεται από το σχεδιασμό του. Τα θέματα τα οποία σχολιάσατε εσείς ε, ήταν κάτι που το περίμενα, αγαπητοί συνάδελφοι. Και νομίζω ότι έχουμε ένα κοινό στόχο, ένα πρόγραμμα που θα λειτουργεί, που θα ε, συνοδεύει τους πολίτες μας σε έναν ε, μεταβαλλόμενο κόσμο. Θα λειτουργήσει όμως αυτό το πρόγραμμα μόνο αν μπορέσουμε να ορίσουμε και τις λεπτομέρειες. Και αυτή είναι η αφετηρία. Φαντάζομαι για εντατικές συζητήσεις και για καλή συνεργασία. Θα έχουμε όμως και έντονες διαπραγματεύσεις. Το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ ε, περιορισμένο. Ελπίζω το αποτέλεσμα πάντως να είναι θετικό. Σας ευχαριστώ όλους για τις σημερινές σας παρεμβάσεις και περιμένω ε, στη... να έχουμε καλή συνεργασία στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε, Αγγέλικα. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών η 7η Σεπτεμβρίου. Αυτή τη βδομάδα λίγη δηλαδή προθεσμία. Επόμενο σημείο θα είναι η συμφωνία με την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Γιατί έχουμε εν μέρη κοινή αρμοδιότητα. Εν μέρη γιατί είμαστε η βασική επιτροπή. Αλλά στα επόμενα βήματα ακολουθούμε με την ΙΜΚΟ. Περνάμε στο σημείο 10 της μερικής διάταξης, στάση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Εισηγητής ε, είναι ο κύριος Κρασνοντεύσκη από την ομάδα ECR. Θα ήθελα να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας αυτής ε, τον Ιούνιο. 13 δις είναι ο προβλεπόμενος προπολογισμό για την έρευνα και ανάπτυξη, συγκεκριμένε ε, δράσεις, ειδικέ δράσεις στον τομέα των επενδύσεων ε, για την άμυνα στην Ευρώπη. Πρόκειται για επενδύσεις και για ενέργειες, δράσεις από διάφορα κράτη-μέλη. Δηλαδή μιλάμε για εταιρικέ σχέσεις μεταξύ κρατών μελών. Ελπίζουμε να δημιουργηθεί έτσι ένας καταλήτης που θα δώσει τόνωση και κίνητρα στη βιομηχανία για να δημιουργηθεί μια επιστημονική βάση ε, στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα αυτό επίσης δεν απευθύνεται μόνο στη βιομηχανία αλλά και στους βιομηχάνους. Έχουμε 500 εκατομμύρια μέχρι στιγμή για τι πρώτε επενδύσει στον τομέα αυτό. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Κρασνοντεύσκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καθορίσατε το, το πλαίσιο της πρότασης αυτής. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό ταμείο για την άμυνα, όπως έχω πει και στο παρελθόν. Έχουμε λειτουργήσει στα πλαίσια της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Έχουμε διαπραγματευτεί διάφορες φάσεις, αναφέρομαι στις διαπραγματεύσεις με την κυρία Γκροσέτ, η οποία είναι ιδιαίτερα δεσμευμένη στον στόχο μας αυτό. Θέλω να υπογραμμίσω αρκετά σημεία στα οποία είχαμε διαξεφιστεί με την Κομισιόν, τα οποία τελικά τα έλαβαν υπόψη τους σε διαφορετικές συναντήσεις με τους ε, Ευρωπαίους νομοθέτες αλλά και με ερευνητικά κέντρα και βεβαίως είναι ανάγκη ακόμη να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα ζητήματα. Θα ήθελα τώρα να θέσω, να την προσοχή σας σε κάποιες τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να αναρωτηθούμε σχετικά με το πώς θα μπορέσουν να συνεργαστούν αυτές οι διαφορετικές επιχειρήσεις, πώς θα λειτουργήσει. Είναι η τροπολογία 42-43 που αναφέρονται σε αυτήν την συνεργασία, σε αυτό το καινούριο μοντέλο συνεργασίας. Μιλάμε εδώ για ένα καινούριο πρόγραμμα, καινοτόμο πρόγραμμα, που δεν θέλουμε να κρατήσουμε το πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε μέχρι στιγμής. Θέλουμε να δώσουμε έμφαση στα προγράμματα που θα αυξήσουν την αυτονομία μας σε σχέση με τρίτες χώρες. Πρέπει επίσης, επίσης να εξακολουθήσουμε να ασχολούμαστε με τα προγράμματα που είναι προγράμματα προτεραιότητας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις προτεραιότητές μας ό,τι αφορά την άμυνα, την ευρωπαϊκή άμυνα. Είμαι πεπισμένο και πιστεύω ότι και οι άλλοι ηγητέ θα συμφωνήσουν μαζί μας ότι είναι ανάγκη να ενδυναμώσουμε τον ρόλο των κρατών μελών. Γιατί τα κράτη-μέλη είναι αυτοί οι οποίοι θα εποφεληθούν από την ανάπτυξη των εργαλείων αυτών χάρη στο πρόγραμμα αυτό. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά στις τροπολογίες αναφέρομαι στα διαφορετικά έγγραφα, τα οποία έχουν συντάξει διάφοροι φορείς, αναφέρονται στην τεχνολογία της άμυνας, σε ευρωπαϊκά πρακτορία αμήνης, αναφέρονται σε τεχνικά ζητήματα Πρόκειται για ένα θεματολόγιο καθολικό. Οι τροπολογίες 39 και 33 ασχολούνται με αυτό το θέμα λεπτομερώς. Επίσης, το ταμείο αυτό της Ευρωπαϊκής Άμυνας θα πρέπει να είναι ευέλικτο. Στην τροπολογία 37 προτείνουμε ότι ένα κομμάτι οικονομικών αποθεμάτων θα μπορούσε να μεταφερθεί από τον πυλώνα αυτό στον δεύτερο πυλώνα. Και τέλος, ένα ζήτημα κάπως αντιφατικό, κάπως ακανθόδες. Αναφέρομαι στο ζήτημα της ειδικής. Εμείς θεωρούμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να μπορεί να διακόψει την χρηματοδότηση ενός προγράμματος αν θεωρεί ότι δεν κινείται προς την σωστή κατεύθυνση από ηθική άποψη είναι οι τροπολογίες 43, 44 και 45 που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό της ηθικής. Εν κατακλείδη, ένα ζήτημα το οποίο έχουμε συζητήσει πολύ στο παρελθόν, πρόκειται για την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση ορισμένων επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από πηγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ζήτημα που είναι συνδεδεμένο με, αυτό το θέμα. Αναφέρομαι εδώ στην τροπολογία 58. Θα ήθελα να, να βγάλουμε από το ταμείο αυτό όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες υπόκειται σε κυρώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να βγάλουμε λοιπόν από τον κατάλογο του Ταμείου αυτού. Πιστεύω ότι η συνεργασία μας θα είναι ιδιαίτερα επικοδομητική. Θα μπορέσουμε να επικεντρωθούμε στο μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και είμαι πεπισμένος ότι οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πρώτη α, παρέμβαση από την κυρία Γκροσέτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά του. Προφανώς και έχουμε κάποιες διαφορές απόψεων, αλλά θέλουμε το Ταμείο αυτό να είναι μια επιτυχία για την Ευρώπη είναι βασικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει προτάσεις θετικές. Είναι η συνέχεια του βιομηχανικού προγράμματος 2019-2020. Δίνει προοπτική στην Ευρώπη της άμυνας πιο φιλόδοξη και με σωστή στήριξη κοινών προγραμμάτων, μικρής ή μεγάλης εμβέλειας. Για μας πιστεύουμε ότι το Ταμείο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί με αποτελεσματικό τρόπο. Θα πρέπει να αποφύγουμε ε, βαρύ, βα, βαριάς μορφής συνεργασίες, ε, περίπλοκες συνεργασίες που θα δημιουργήσουν καθυστερήσεις. Πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα ε, και έτσι θα μπορέσουμε να διασώσουμε την βιομηχανία μας. Ο προϋπολογισμός των 13 δις ανάμεσα στην έρευνα και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων είναι το ελάχιστο δυνατό όταν βλέπουμε τα διακυβεύματα και τις προκλήσεις που υπάρχουν έτσι ώστε να καταστεί η Ένωση ανεξάρτητη. Ε, Σύμφωνο απόλυτα με την πρόταση ε, το 5% του προϋπολογισμού για τις λεγόμενες τεχνολογίες ρήξης. Είναι το ελάχιστο και όχι όριο ανώτατο. Πρέπει να δούμε και τις μικρομεσές που χρειάζονται τη βοήθεια αυτή για να λειτουργήσουν στα πλαίσια των κοινών προγραμμάτων. Πρέπει λοιπόν εμείς να βοηθήσουμε τις μικρομεσές χωρίς διακρίσεις με πόνους για τις μικρομεσαίες που δεν βρίσκονται στο κράτος μέλος της αρχικής επιχείρησης όπως το κάναμε το 1920 για το πρόγραμμα 1920. Τώρα, σχετικά με το δεοντολογικό θέμα που αναφέρεται στο άρθρο 7, η ιδέα είναι καλή επί της ουσίας, δημιουργεί όμως μια νομική ανασφάλεια σε σχέση με τι σημαίνει ένα δεοντολογικά σωστό πρόγραμμα, και στην ικανότητα να προχωράμε σε νέου είδους προγράμματα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται εκ των προτέρων αυτός ο δεοντολογικός έλεγχος, αν για δεοντολογικούς λόγους το πρόγραμμα δεν είναι επιλέξιμο, πρέπει να το γνωρίζουμε εξ αρχής. Τώρα για τα κριτήρια επιλεξιμότητας υπάρχουν αρκετές θετικές προτάσεις, έχουμε ένα ισορροπημένο κείμενο, Έχουμε κάποιες ε, ρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν για να διασφαλιστεί ο σωστός χαρακτήρας του ευρωπαϊκού χαρακτήρα της προσπάθειας για να ενισχυθεί η στρατηγική ανεξαρτησία της Ένωσης και ε, αν χρειάζονται εμπόδια και φράγματα σε ένα τέτοιο στρατηγικό τομέα θα πρέπει να τα για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας. Καλό θα είναι να τα εναρμονίσουμε ανάμεσα στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρήζει περισσότερης επεξεργασίας. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία μου φαίνονται τα πιο σημαντικά για την ομάδα μου. Θα στηρίξουμε την γρήγορη επεξεργασία του κανονισμού αυτού μέσω τροπολογιών. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά και εγώ είμαι υπέρ μιας ευρωπαϊκής άμυνας. Πρέπει όμως να επαγρυπνούμε σε ό,τι αφορά τα κείμενα τα οποία προτείνει η Κομισιόν και το κείμενο της ηγητού εδώ. Υπάρχουν κάποιε διαφωνίε και σε ό,τι αφορά τον τύπο και σε ό,τι αφορά την ουσία. Σε ό,τι αφορά τον τύπο, τη διαδικασία δηλαδή, καταλαβαίνουμε γιατί ε, υπάρχει αυτή η βιάση, να έχουμε δηλαδή μια συμφωνία για αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, που σίγουρα θα είναι ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και στο σημερινό διεθνές γεωπολιτικό πλαίσιο, είναι κάτι δικαιολογημένο, όμως δεν θα ήταν, θα ήταν μάλλον παρακινδυνεμένο να πάμε στα τυφλά λίγο με αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, για αυτό το πρόγραμμα και για άλλα μέχρι το τέλος της θητείας εφόσον δεν έχουμε ακόμη συμφωνήσει για το πολιτέ μεσορμικό πλαίσιο και υπάρχουν ακόμη μεγάλες ε, αποκλήσει μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ναι, με, πρέπει να υποστηρίξουμε την ευρωπαϊκή πολιτική άμυνα ε, και θα πρέπει να ενταχθεί ε, στο πολιτές σωμικό πλαίσιο, ο προβλησμός αυτής της πολιτικής δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρος άλλων πολιτικών. Όμως δεν έχουμε καμιά ορατότητα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται μέχρι το τέλος της θητείας και αν δούμε ποια είναι η θέση κάποιων κρατών μελών μας δημιουργεί προσωπικά εμένα τουλάχιστον μεγαλύτερες ακόμη αμφιβολίες που ε, είπαμε, ε, είδαμε τι λένε τα ε, κράτη. Ψηφίστε σε αυτό και αφήστε μας εμάς ήσυχους για όλα τα άλλα. Ποια είναι όλα τα άλλα. Η ουσία. Και έρχομαι στην ουσία. Έχουμε την πρώτη Κομισιόν ε, που περιλαμβάνει και πολλά στοιχεία από την έκθεση Γκροστέτ και ο εισηγητής και συμφωνώ, αλλά υπάρχουν και πραγματικές αποκλήσεις κατά τη δική μου άποψη και την άποψη της ομάδας μου. Άρθρο 10 πρώτα απ' όλα. Επιλέξουμε οντότητες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι συμβιβασμός, όμως εγώ εξακολουθώ να έχω τις αμφιβολίες μου. επειδή θα καλύψει μεγάλο μέρος της κατάστασης του 2020. θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι σε κάποια κράτη υπάρχει ακόμα η μη ευρωπαϊκή συνιστόσα που είναι σημαντική, αλλά αυτό μπορεί στο μέλλον να αλλάξει. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ευρωπαϊκές κοινοπραξίες στο μέλλον. Στο ίδιο πνεύμα. Θα πρέπει τα κριτήρια ανάθεσης ε, να αναβαθμιστούν, να ενισχυθούν σε σχέση με την τεχνολογία που μπορεί να δημιουργήσει έναν άρρητο κύκλο σε κάποια συγκεκριμένη χώρα. Θα πρέπει να υπάρξει προσέγγιση της χρηματοδότησης ε, όμως με τους στόχους, όπως είναι η ΠΕΣΚΟ για παράδειγμα. Άρθρο 7 τώρα και ηθικά θέματα, το ηθικό σκέλος. Δημόσια κονδύλια χρηματοδοτούν αυτό το πρόβλημα. Οπότε τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να κοιταχθούν στον καθρέφτη και θα πρέπει να ενισχυθεί αυτό με δύο τρόπους. Οι εκπρόσωποι του λαού, εμείς δηλαδή, θα πρέπει να μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τους ε, ηθικούς και άλλους εμπειρογνώμονες και να δούμε τα στήματα αυτά όχι μόνο υπό το πρίσμα της τεχνολογίας αλλά και του δυνητικού πλαισίου χρήσης αυτών των τεχνολογιών. Φυσικά και δεν είναι απαγορευμένο να πολλούμε στην ε, Σαουδική Αραβία όπλα, αλλά ε, δεν πρέπει να ε, δούμε τι γίνεται με αυτά τα όπλα που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στην Ιεμένη. Ε, γι' αυτό θέλω να υπάρχει αυτή η διάσταση στην ε, έκθεση. Και έχουμε τέλος και το άρθρο 29 για τους εμπειρογνώμονες. Δεν μπορούμε νομίζω να υποστηρίξουμε ότι θα πρέπει να μείνει κρυφός ο κατάλογος. Εμείς θέλουμε αντίθετα περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη δημοκρατία. Τέλος χρηματοδότηση προγραμμάτων αμυντικών εξοπλισμών, μεγαλύτερη πελατειακή βάση είναι καλύτερο από το να αναζητούμε μόνο τις εξαγωγές εκτός Ευρώπης. Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε το business as usual με πρόσθετη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αυτή η προσέγγιση που σας αναφέρω μου φαίνεται πολύ πιο λογική. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο, λέει ο πρόεδρος. Για το άλλο έχει το λόγο ο κύριος Λεκουέτς. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Μετά την προηγούμενη έκθεση συνεχίζουμε. Πρόκειται για μια έκθεση πιο σημαντική σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον η εισηγητή για αυτή την εξαιρετική δουλειά με την οποία συμφωνούμε σε μεγάλο μέρος. Κάποια σημεία όμως που έχουμε επιφυλάξεις. Καταλαβαίνω τι λέει ο Εντουάχα σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαι αρκετά ικανοποιημένος με τα νούμερα που παρουσιάστηκαν. Είναι ένα ζήτημα που πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Μπορούμε να συζητήσουμε διάφορα σημεία σε ό,τι αφορά ας πούμε, τις συγκεκριμένες παραμέτρους του προϋπολογισμού. Αλλά αυτή η συζήτηση είναι πιο ευρεία. Θέλω να μην μακρηγορήσω. Έχω και εγώ αυτό το, το ζήτημα ε, επιλεξιμότητας. Είναι ίσως περίεργο να, να πούμε ότι πρόκειται για ένα τεχνικό θέμα. Είναι ένα θέμα ευρωπαϊκής αυτονομίας. Σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα, είμαι ιδιαίτερα δύσπιστος σε ό,τι αφορά την επιλογή οντοτήτων που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που έχουν αναπτύξει την τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία. Δεν έχω δει εταιρείε που να βρίσκονται στις Ηνωμένε Πολιτείε ή στη Γαλλία να συνεργάζονται με κινέζικες εταιρείε. Ίσως είμαι πολύ δύσπιστος, ίσως είμαι πολύ αφελής σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των συνεργασιών. Μπορεί να δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση των επενδύσεων, όπως αυτά που ανέφερε και ο Έντουαρτ Μαχτάν, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα εξαγωγών. εξαγωγών. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος των εξαγωγών αν αγοράζει κανείς ένα μαχαίρι πρέπει να, να ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιηθεί. Ξέρουμε ε, επίσης ότι οι εξαγωγές είναι αυτές οι οποίες ε, οδηγούν και την παραγωγή. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να συγχαρώ την έκθεση σε ό,τι αφορά τον τομέα της έρευνας. Πιστεύω ότι η Γκροστέτ ε, ήταν κέρια τα, τα σημεία που έθιξε. Σε ό,τι αφορά και την ε, τεχνολογία στη διάθεση των πολιτών, θα πρότεινα να περάσουμε από το 5% στο 10% εγώ προσωπικά, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό για την έρευνα πιστεύω ότι θα ήταν αντιπαραγωγικό να αντιταθούμε σε αυτό το κομμάτι του προπολογισμού για την έρευνα. Υπάρχουν και άλλα σχόλια, πιο συγκεκριμένα, αλλά έχουμε την εντύπωση ότι συμφωνούμε σε γενικές γραμμές με τον εισηγητή. Υπάρχουν κάποιες διαφωνίες. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να, να συμφωνήσουμε. και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις. Γιατί, όπως σας είπα και προηγουμένως, θεωρώ ότι είναι ένα κέριο ζήτημα ευρωπαϊκής οικονομίας. Ε, αυτονομίας, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Σιλικιώτη, από την ΚΟΕ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ξεκάθαρο πως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας αποτελεί μέρο του ευρύτερου σχεδίου για την οικοδόμηση τη Στρατιωτικής Ένωσης. Ε, μέσω βεβαίω και του στόχου για ενίσχυση τη στρατιωτική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θέση που εμεί ε, υποστηρίζεται και από τον εισηγητή τη έκθεση. Ε, ο μίσο ομάδα είμαστε ενάντια σε τέτοιε ε, επικίνδυνε πολιτικέ και επικίνδυνο εγχείρημα, ιδιαίτερα σήμερα σε έναν κόσμο που μαστίζεται με πάρα πολλού περιφερειακού πολέμου και η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται τι αρνητικέ συνέπειε αυτών των πολέμων, όπω των πολέμων που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση που έχει καταθέσει να γίνουν επενδύσει στην άμυνα ύψου 13 δισεκατομμυρίων για την περίοδο 21-27. Ειδικότερα προτείνεται και η δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνα για την υποστήριξη επενδύσεων στην άπτυξη αμυντικών προϊόντων. Εμεί τα ονομάζουμε επιθετικά προϊόντα και όχι αμυντικά προϊόντα. Και τεχνολογιών για την πρόθεση τη αγορά και συντήρηση αμυντικών εξοπλισμών από τα κράτη-μέλη. Μέσω αυτή τη ε, επένδυση η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύσει στον πόλεμο. Επενδύει στι εξαγωγέ όπλων ευρωπαϊκών χωρών, τη ε, ευρωπαϊκή στρατηγική βιομηχανία, ειδικότερα σε ε, ζώνε όπω είναι η Μέση Ανατολή που είναι πολύ κρίσιμη. Πρέπει να πω ότι το 2016 το 1 τέταρτο των εξαγωγών όπλων τη Γερμανία ήταν στη Μέση Ανατολή. Σε μια περιοχή που έχουμε τον εμφύλιο πόλεμο στην Ιεμένη, στη Συρία, τους καθημερινούς πολέμους με τις χιλιάδες ε, ε θανάτους και τα εκατομμύρια πρόσφυγες ε, που υποφέρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αυτού. Το άλλο στοιχείο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η πρόταση της Επιτροπής παραβιάζει εξόφθαλμα το, τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραβιάζει το άρθρο 41, την παράγραφο 2 της συνθήκης της Ένωσης, που αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι δαπάνες που προκύπτουν από επιχειρήσεις που έχουν στρατιωτικές ή αμυντικές συνέπειες δεν πρέπει να χρώνονται στον προπολογισμό τη Ένωση. Αυτό λέει η συνθήκη και μέσω αυτή τη δημιουργία αυτού του ταμείου ε, και αυτή τη επένδυση ε, παραβιάζεται αυτή η συνθήκη και είναι αυτό που δυστυχώ επιχειρείται σήμερα. Ω ε, QNGL θα καταθέσουμε τροπολογία για συνολική απόρριψη τη πρόταση που κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία δηλαδή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας Εμεί ζητάμε να αξιοποιηθεί αυτό το κοντίνι των 13 δισεκατομμυρίων για την πρόθεση τη ανάπτυξη, ιδιαίτερα στα κράτη και στι περιοχέ που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, στη βάση των αγκών τη κοινωνία. Ή αν η Ένωση σέβεται τι διακριμένε αρχέ τη, οφείλει να πάψει να επενδύσει στου πολέμου και αντί αυτού να επενδύσει εκεί που χρειάζεται η ανάπτυξη και να καταστεί πυλώνα ειρήνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Εκ μέρου του e ΙΕΝΕΦ. Κυρία Τεσεβαλή, έχει το, το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο στόχος ε, να ευνοηθεί η αριστεία της Ευρωπαϊκή ε, αμυντικής βιομηχανίας ε, είναι θετικός όπως και η προμήθεια ε, εξοπλισμού από χώρες της Ένωσης και όχι τρίτες χώρες. Όμως στόχος εδώ είναι να υπάρξει αλληλεξάρτηση των ε, στρατών και των αμυντικών βιομηχανιών μας και όχι η μεγαλύτερη αυτονομία. Και αυτό ε, υπέρ μιας μη θεμητής ευρωπαϊκής άμυνας και γι' αυτό είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε κάποιες παρατηρήσεις οι συνδεδεμένε χώρε, μεταξύ αυτών και η Τουρκία. Ε, δίνεται σημασία σε αυτό. Υπάρχουν τροπολογίε 8, 65 και 85. Ε, δεν είναι, επαρκή, είναι όμως επαρκής. Έχουμε Επίσης, μια διαφορετική μεταχείριση στη Ρωσία, Εμέσω εμέσως ε, στην τροπολογία 11. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κάποια εξαίρεση. Είπαμε ότι είναι πολύ καλό το ΠΕΣΚΟ, έχουμε την 72 που ενισχύει αυτή την συνεργασία. Όμως ε, μιλάμε για υπαγωγή στους στόχους του ΝΑΤΟ μέσα στις τροπολογίες 18. Και τέλος, για την 73 τροπολογία, στόχος είναι να μην δώσει ε, σημασία σε χώρες όπως είναι η Γαλλία. Ε, όποια και αν είναι η πολιτική που ακολουθείται, πρέπει να ξέρουμε ότι φορολογούμενοι των χωρών είναι αυτοί που πληρώνουν. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Κύριο κύριος Γκάιερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Καταρχάς, θέλω να πω ότι δεν είμαι σκιώδης εισηγητής για την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, άρα λαμβάνω προσωπικά το λόγο ως ε, Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης, διότι θεωρώ ότι στην ομάδα μας Υπάρχουν κάποιες ε, διαφωνίες ε, μικρές ό,τι αφορά αυτή την ε, πολιτική και αυτό το τάμε Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω κάποια σημεία με τα οποία έχουμε σημαντικά προβλήματα. Κατά την άποψή μου, ξεκινάμε με μια πολύ μικρή ουσιαστικά συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε την ηθική αξιολόγηση λέμε μόνο κατόπιν σε στάσεως της Κομισιόν. Ξεκινάμε δηλαδή ήδη από εκεί αφήνοντας εκτός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και μιλάμε για εξαγωγές ε, αμυντικών προϊόντων. Αυτό είναι καυτή πατάτα στη Γερμανία και είναι ένα πάρα πολύ ε, σημαντικό ζήτημα το οποίο το, μας δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες να υπάρχουν αυτοί οι κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα ε, εγκρίνουν και που είναι πολύ πιο χαλαροί αυτοί οι κανόνες από ό,τι θα θέλαμε. Και γνωρίζουμε και από την γερμανική πολιτική ότι ε, μπορεί να προκύψει με την ε, νομιτικό εξοπλισμό κάποιων χωρών. Και αυτό, αυτά τα προβλήματα δεν προκύπτουν μόνο από τις εξαγωγές αλλά και από άλλα ζητήματα. Ε, υπάρχουν ε, στρατηγικά ζητήματα που πρέπει να αξιολογούνται σε κάθε περίπτωση. Και από την άλλη πλευρά έχουμε το θέμα της χρηματοδότησης των ε, στόχων ε, και από ποιους άλλους ε, τομείς θα μπορούσαν να προέλθουν τα κονδύλια. Και εκεί βρίσκω και εγώ άλλο πρόβλημα. Θέλουμε να έχουμε ένωση και από κοινού χρησιμοποίηση δυνατοτήτων. Αυτό είναι καλό μένα. Από την άλλη πλευρά πρέπει να ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρξουν απώλειες θέσεων πού θέλουμε να χαθούν αυτές, ε, ε, θέλουμε να έχουμε ένα ή δύο μόνο ή θωρακισμένων ή 13. υπάρχουν κάποια, κάποια απαρχιωμένα άρματα μας. Τι θα γίνει και τι θα γίνει με την μετατροπή. Είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Και ε, έχουμε ασκήσει και ασκούμε έντονη κριτική και σε αυτό το πεδίο. Επίσης, ρητός στόχος, ε, είναι ε, οι εθνικές αμυντικές δαπάνες. Αυτό για μας είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχθούμε. Επίσης θετικό θα ήταν να είχαμε έναν, έναν ισχυρό ε, ερευνητικό τομέα για να παραμείνουμε ανταγωνιστικό, αλλά αυτό το παράθυρο στην έρευνα. Νομίζω με αυτή τη στοχοθέτηση ε, δεν πρόκειται να δημιουργηθεί. Σε ό,τι δεν αφορά τη νομική βάση, δεν είμαστε ικανοποιημένοι και δεν είναι πιστική η πρόταση της Κομισιόν. Στην τελευταία ε, συζήτηση ακούσαμε ότι η στρατηγική αυτονομία δεν μπορεί να είναι θέμα. Το είπε όμως και ο συνάδελφος από την αριστερά. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα με συμβατότητα με τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Ναι ή όχι. Αν υπάρχει στρατηγική αυτονομία. Ε, υπάρχει. Ε, και πού λέγεται στις συνθήκες για τις αμυντικές ε, βιομηχανίες και την ε, στρατηγική αυτονομία σε σχέση πάντα με, τις αμυντικές, με τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την έκθεση που μας παρουσίασε, η οποία έκθεσή του στηρίζει και την πρόταση της Κομισιόν. Υπάρχουν ζητήματα που θα πρέπει να επανεξετάσουμε, αλλά σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με τη θέση του εισηγητή. Στην παρούσα φάση θέλω να εφιστήσω την προσοχή σας σε δύο σημεία. Το πρώτο έχει να κάνει με την πιθανή συμμετοχή τρίτων χωρών. Η πρόταση της Κομισιόν αντανακλά αυτά τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί και έχουν γίνει αποδεκτά από το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και στα πλαίσια του προϋπολογισμού α, όπου και συζητήσαμε την α, ιδέα του να εστιάσουμε σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις των κρατών μελών και να μην χρηματοδοτούμε επιχειρήσεις τρίτων χωρών ή που βρίσκονται κατεστημένες σε τρίτες χώρες. Σε κανένα τρόπο δεν μπορεί μια επιχείρηση τρίτης χώρας να υποφελείται από κοινοτικά επιδόματα. Αλλά επιχειρήσεις που στηρίζονται από τρίτες χώρες θα μπορούσαν ίσως να επωφεληθούν από κοινοτική χρηματοδότηση. Επιμένουμε σε αυτήν την ευελιξία που πιστεύουμε ότι μπορεί να αποβεί επωφελής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπογραμμίζω ότι πρόκειται για πολύ ειδικέ περιπτώσεις, ούτως ώστε να μπορέσει η Κομισιό να έχει μια ισορροπία για αυτήν την πιθανή συνεργασία. Το δεύτερο σημείο που θέλω εντάχει να θίξω έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση του προγράμματος. Είναι σημαντικό να σας πενθυμίσω ότι πρόκειται για ένα κοινοτικό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης βιομηχανικής στα πλαίσια της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τις πολιτικές της άμυνας. Έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Και αυτός είναι ο λόγος που καθιστά σημαντικότητα το να παραμείνουμε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, να υπάρχει έλεγχος από τις αρχές του προϋπολογισμού. Η επιτροπολογία είναι πάρα πολύ σημαντική για την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας, κυρίως σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις προτεραιότητες έτσι όπως έχουν προκαθοριστεί. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας διάφορες ατιφάσεις, να μην μπερδεύουμε το κοινοτικό πλαίσιο με το διακυβερνητικό πλαίσιο. Είναι ανάγκη να διατηρήσουμε την ισορροπία αυτή που θα μας επιτρέψει να επωφεληθούμε στο μέγιστο από την συνεργασία των διαφορών φορέων. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και είμαι βεβαίως στην α, διάθεση των εισηγητών. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον εισηγητή, ούτως ώστε να μπορέσει να συνοψίσει λίγο τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση που προηγήθηκε είναι πολλά υποσχόμενη. Δεν νομίζω ότι θα ε, βαρεθούμε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει στο μέλλον. Υπάρχουν θέματα όπως ε, η επιλογή των προγραμμάτων, όπως η συμμετοχή τρίτων χωρών. Είναι όλα θέματα τα οποία από ό,τι φαίνεται θα προκαλέσουν πολλές συζητήσει. Υπάρχουν και γενικότερες απορίες αλλά ε, θα συγκεντρώσω την προσοχή μου ε, στο θέμα της συμμετοχής των τρίτων χωρών. Ακούστηκαν κάποια επιχειρήματα, ακούστηκαν θέματα όπως η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το, ε, υπάρχουν πολλοί εμπειρογνώμονες μεταξύ των οποίων και Γάλλοι, πιστεύουν ότι το ΝΑΤΟ είναι αυτό το οποίο μέχρι τώρα ουσιαστικά διασφαλίζει την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε οποιαδήποτε αλλαγή εδώ θα ήταν, θα έλεγα, επαναστατική. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να προβλέψουμε λοιπόν την συμμετοχή των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αλλά να συνεργαστούμε και με τη Μεγάλη Βρετανία και με τις Ηνωμένε Πολιτείες και μετά το Brexit θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργάζεται σε στρατηγικό επίπεδο με το Ηνωμένο Βασίλειο. Φυσικά υπάρχουν ορισμένες αμφιβολίες. Ο Γερμανός συνάδελφος είπε ότι το κόμμα του είναι κατά της αύξησης των δαπανών για το θέμα της άμυνας. Ε, το κόμμα του όμως, όχι η κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει. Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία φυσικά τίθενται και από ό,τι φαίνεται εδώ ε, πουλήθηκαν ε, πολλά όπλα γερμανικής προέλευσης στις ε, περιοχές τις οποίες υπάρχουν συγκρούσεις χένουσες αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά δείχνουν ότι ε, υπάρχουν αρκετά εμπόδια, υπάρχουν αρκετά αγκάθια στο πρόγραμμα αυτό. Θα πρέπει να καταστήσουμε το πρόγραμμα ε, ιδιαίτερα αποτελεσματικό, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε ε, την αμυντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ταυτόχρονα να σεβαστούμε τις αρχές ε, που ισχύουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους ε, τους σκιώδεις ε, και τους υπόλοιπους ομιλητές. Η προθεσμία κατάθεσης των τροπολογιών είναι η 12η Σεπτεμβρίου και οι υπόλοιπες προθεσμίες θα καθοριστούν σε εύθετο χρόνο. Περνάμε αμέσως στο σημείο 11. Η κυρία Γιούρκουνεν θα μας παρουσιάσει, θα μας δώσει πληροφορίες σχετικά με την αποστολή μας στην Νορβηγία. Α, η κυρία Γιούρκουνεν είναι απούσα, οπότε αναβάλλεται το θέμα αυτό για τις 24 Σεπτεμβρίου. Έχετε κάποιες παρατηρήσεις γύρω από όλα αυτά. Όχι, τότε θα διακόψουμε και θα συναντηθούμε στις 19 Σεπτεμβρίου στην όμορφη πόλη του Στρασβούργου. Σε μία εβδομάδα, λέει ο πρόεδρος, 5.30 το απόγευμα, πολύ σημαντική συνάντηση. Δεν θα έχουμε πολύ χρόνο Οπότε παρακαλώ να είστε εκεί εγκαίρως. Ευχαριστώ πολύ. Θα συναντηθούμε λοιπόν σε μία εβδομάδα. Γεια σας.